Good afternoon. Uh, Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι της Επιτροπής Ελίμπε και ΕΚΟΝ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτή την κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών. Όπως ξέρετε, η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε πώς σήμερα θα συζητήσουμε την οδηγία κατά του ξεπλήματος ε, χρήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα 51. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο μας επιτροπές θα συνεργαστούν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και με χαρά καλωσορίζω την κυρία Άστρη Λούλιν, την συμπρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι η πρόεδρος της Επιτροπής Οίκων, ούτε καν η αντιπρόεδρος, αλλά εξαφανίστηκαν όλοι. Έτσι λοιπόν το γυρεότερο μέρος, μέλος του Ευρωκοινοβουλίου έπρεπε να έρθει. Για να μιλήσω και γαλλικά, χαίρομαι πάρα πολύ βέβαια που έχω το καθήκον αυτό λάβει γιατί το θέμα είναι άκρο ενδιαφέρον, δηλαδή η αποτροπή της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ε, για την ομοποίηση εσόδων παράνομης δραστηριότητας και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και θα ήθελα να συγχαρώ τους τέσσερις εισηγητές, συνεισηγητές Δύο είναι, αλλά τέλος πάντων για τις εκθέσεις που εκπώνησαν, που είναι πολύ καλές και μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε. Θα δώσω ευθύς αμέσως το λόγο στον εισηγητή Κάρινς. Πέντε λεπτά έχει στη διάθεσή του. Τέσσερα 47 θέλατε, αλλά θα, θα σας δώσω 4,5. Ωραία, θα τα καταφέρω. Αγαπητοί πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς εδώ στην αίθουσα με τον εκπεφρασμένο στόχο της ε, οδηγίας μας βρίσκει όλους ε, σύμφωνους. Δηλαδή, για την φοροδιαφυγή και την ε, νομοποίηση εσόδων πάνω στις δραστηριότητες, να τα δυσκολεύουμε στο δυνατόν περισσότερο, απομακρύνοντας ε, τα εγκληματικά δίκτυα και τις εγκληματικές δραστηριότητε, ως το δυνατόν περισσότερο. Θα ήθελα να σας πω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Εμένα τουλάχιστον προξένησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η κυρία Σαρτζεντίνη ανέλαβε μαζί με μένα το πολύ ενδιαφέρον καθήκον να συντάξουμε μία έκθεση η οποία προέρχεται από δύο διαφορετικές ε, επιτροπές αλλά και από δύο διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Ξέρετε ότι ως μέλη διαφορετικών πολιτικών ομάδων δέχεται να έχουμε διαφορετικές απόψεις για το τι είναι σημαντικό, για το που πρέπει να δώσουμε έμφαση και η κυρία Σαντζετίνη και εγώ δαπανίσαμε αρκετό χρόνο πάνω σε αυτό και το προϊόν τη κοινή μα δουλειά είναι κοινή μα συμφωνία, ένα τάγραφο που σα υποβάλλουμε. Κάναμε ένα ενδιαφέρον ταξίδι. Η συζήτηση έχει γίνει βέβαια σε πολύ μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι έχουμε καταλήξει για κάποια θέματα και σε πολύ καλούς συμβιβασμού. Θα ήθελα να αναφέρω τέσσερα θέματα. Η συνεισηγήτριά μου φαντάζομαι θα αναφέρει τα ίδια θέματα και θα επεκταθεί πάνω σε αυτά. Το πρώτο, κάτι που δεν προερχόταν αρχικά από την Κομισιόν, είναι πληροφορίες ε, για το δικαιούχο ιδιοκτησίας. Πληροφορίες ιδιοκτησίας για το δικαιούχο. Είναι καλό να καταπολεμήσουμε την, ε, το ξέπλυμα χρήματος εάν έχουμε ένα μητρό που έχουμε αυτούς τους δικαιούχους μέσα. Στην Λιτωνία, για παράδειγμα, έχουμε αυτό το μοντέλο, έχουμε την αποκάλυψη των πληροφοριών για τα στοιχεία για την ιδιοκτησία οποιασδήποτε επιχείρηση. Αλλά μπορεί να δει κανεί ότι το, ο John Doe, για παράδειγμα, έχει 49% και κάποια άλλη επιχείρηση μέτρα σε ένα άλλο κράτο έχει το 51%. Αυτό μπορεί να το δει κανεί, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο κρύβεται πίσω από το 51%. Γιατί το άλλο κράτος μέλος ε, ενδεχομένω να μην διαθέτει τις πληροφορίες αυτές σε ένα δημόσιο μητρό. Να μην τα ξεκάθαρα τα πράγματα δηλαδή στο άλλο κράτος μέλος. Άρα η ιδέα μας είναι αυτά τα μητρώα να, να τα ανοίξουμε και να τα διασυνδέσουμε το ένα με το άλλο. Ενδιαφερόμενες αρχές, φορολογικές, αστυνομικές και άλλες, τράπεζες επίσης, υπόχρες οντότητες να μπορούν να δουν ποιος είναι πίσω από αυτή την εταιρεία, ώστε οι συναλλαγές ε, να είναι δηλωμένες και να πληρώνεται και ο φόρος εκεί που πρέπει. Οι συζητήσεις που είχαμε δεν αφορούσαν τόσο πολύ το κατά πόσο θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο μητρό, αλλά το θέμα μας ήταν το επίπεδο της διαφάνειας. Εγώ νιώθω άνετα με ένα επίπεδο διαφάνειας που σημαίνει ότι υπόχρεες οντότητες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του Μητρό και τα κράτη-μέλη από εκεί πέρα θα επιλέγουν πόσο θα δημοσιοποιήσουν το Μητρό αυτό. Για τα θέματα της φοροδιαφυγής, ακριβώς αυτές οι υπόχρεες οντότητες που πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και εάν είναι δημόσιο το Μητρό, ουσιαστικά δεν καλύπτονται εντελώ ε, το θέμα. Μπορεί να βοηθήσει δηλαδή την ε, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά επειδή υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση, θα μπορούσαν να στοχεύονται πιο εύκολα ορισμένα θύματα, άρα οι εγκληματικέ δραστηριότητε να ευνοηθούν. Για τα εκτεθειμένα άτομα, το σημείο 2, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να συνταχθεί ή να υποβληθεί, αν θέλετε, ένα κατάλογο από τα κράτη-μέλη που γνωρίζουν και είναι αυτά πολιτικώς εκτεθειμένα άτομα, βέβαια χρειάζεται ένα συντονιστεί. Και με τον Επίτροπο είχα κάποιε συζητήσει, υπάρχουν κάποιε επιφυλάξει από ό,τι κατάλαβα για το θέμα αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο τρόπο ε, να συντονίσουμε έναν τέτοιο νέο κατάλογο. Θα μα βοηθήσει αυτό και στην συγκεκριμένη προσπαθία. Τρίτο, αξιολόγηση κινδύνων. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση του ξεπλήματο χρήματο να βάλουμε τις προσπάθειές μας εκεί που υπάρχουν κίνδυνοι και να δούμε συγκεκριμένα ποιοι είναι οι προβληματικοί τομείς. Η Κομισιόν θα πρέπει να αναλάβει το διακρατικό επίπεδο, την ε, ευρωπαϊκή δηλαδή αξιόλογηση κινδύνου. Τέταρτο, προστασία δεδομένων. Και γι' αυτό συζητήσαμε αρκετά οι δύο συνεισηγητές. Σίγουρα θα πρέπει η νομοθεσία αυτή να δημιουργεί ασφάλεια για την βεβαιότητα, για την ε, επιχειρηματική κοινότητα. Στόχος της οδηγίας είναι η καταπολέμηση του και η προστασία των δεδομένων καλύπτεται από άλλε οδηγίες, πράγματι. Είναι ένα παράγωγο, αν θέλετε, ένα εγωπροϊόν αυτή τη οδηγία. Εμεί έχουμε κάνει αναφορέ σε αρκετέ άλλε οδηγίε. Δεν είναι αντικείμενο η προσέγγιση αυτό καθ' αυτό ως θέμα, αλλά δεν θα πρέπει να τους βοηθάει τους εγκληματίες. Είναι ισορροπημένη πρόταση γενικά, πιστεύω, και ελπίζω να συμφωνήσετε όλοι από της Γενικής Αρχής. Το πόσο τώρα ανοιχτές ή κλειστές θα πρέπει να είναι αυτές οι πληροφορίες, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και γιατί. Uh, and with that, I took my 4.5 minutes and I made it probably into more. Ελπίζω να έχετε κατανοήσει αυτά που είπα και είμαι στη διάθεσή σας. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κάρινς, κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Ναι, ναι, σήμερα θα μιλήσω Ολλανδικά. Ο συνάδελφος και συνεισηγητής κύριος Κάρινς ήδη ανέφερε πολλά σημαντικά θέματα και θα επαναλάβω ορισμένα από αυτά, μπαίνοντας σε περισσότερες λεπτομέρειες από τη δική μου οπτική γωνία. Καταρχάς όσον αφορά το μητρό ιδιοκτησίας των δικαιούχων. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο ακόμα και η Κομισιόν προτείνει οι ίδιες οι εταιρείε να έχουν την υποχρέωση να γνωρίζουν ποιοι είναι οι μέτοχοί τους, ποιοι είναι οι δικαιούχοι τους. Η αλήθεια είναι πως ε, η πρόταση μέχρι τώρα είναι αναπαρκής και Πιστεύουμε πως ένα μητρό είναι πολύ καλύτερη λύση, ένα μητρό που θα είναι προσβάσιμο στο κοινό. Εγώ θα υποβάλω αντίστοιχες ετροπολογίες και είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα, τα μέσα ενημέρωση, του δημοσιογράφου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε τι ακριβώς ε, συμβαίνει. Ένα ανοιχτό μητρό δεν θα είναι βέβαια κάτι εύκολο αλλά πιστεύω πως έχουμε μεγάλη στήριξη. Δεύτερη άποψη, προστασία δεδομένων. Σε περίπτωση που αλλάζει κάποιο σύστημα, από, την, ε, από τις βασικές αρχές λειτουργίες του μέχρι τις λεπτομέρειες πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε η προστασία δεδομένων να εγγυάται. Και εμείς ως Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να διεξαχθούν οι κατάλληλες εκτιμήσεις κινδύνου έτσι ώστε να έχουμε ένα σημείο εκκίνησης, μια φετηρία, μια βάση αυτών των ε, συστημάτων. Όχι μόνο για το ποιοι κρύβονται πίσω από τους δικαιούχους, αλλά για το τι ακριβώς ε, συμβαίνει. Αυτό είναι σημαντικό και για τους ε, πελάτες και για τις επιχειρήσεις και για ε, τις δημόσιες αρχές. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ειδική αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία θα ελέγχει εάν οι διαδικασίες διεξάγονται έτσι όπως θα έπρεπε. Εμείς ε, θεωρούμε για παράδειγμα πως ένας πελάτης πρέπει να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες ε, και να μπορεί να απευθυνθεί στην κατάλληλη υπηρεσία. και σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα μέσα για να οδηγηθεί στην δικαιοσύνη και να καλύψουμε οποιαδήποτε νομικά κενά μπορούν να προκύψουν σχετικά με την ε, προστασία των δεδομένων. Τώρα, τα νομικά πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να είναι είτε μέλη του Κοινοβουλίου, είτε απλή θνητοί όπως εσείς και εγώ. Από τα η εταιρεία World Check είναι μια βρετανική εταιρεία η οποία πουλά προσωπικά δεδομένα των πελατών της και με αυτόν τον τρόπο κερδίζει χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ και οι συνεισηγητές μου προτείνουμε κάθε κράτος μέλος να είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την κατάρτιση των ε, του καταλόγου των δικαιούχων. Ένας κατάλογος στον οποίο θα προσταφερούνται ονόματα. Αυτό φυσικά δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά είναι μια καλή αρχή. Τέλος, να πω ότι η νομοθεσία σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος ε, έχει το σκοπό να συλλάβει τους εγκληματίες. Πολύ συχνά όμως έχει και παρενέργειες. Δηλαδή, εάν εμεί κάνουμε εξαιρετικά δύσκολο ή αδύνατο να μεταφέρει το κεφάλαιο σε χώρες με πολύ κακή φήμη, τότε θα βρουν άλλες οδούς. Η διασπορά και οι απόδημοι στην Ευρώπη θα βρουν άλλους τρόπους για να μεταφέρουν ε, χρήματα παράνομα. Στη Σομαλία, για παράδειγμα, λόγω της κατάστασης, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις είχαν πρόβλημα να στείλουν βοήθεια εκεί, λόγω της ε, απαγόρευσης σχετικά με την ε, κατά με την απαγόρευση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Και πιστεύω πως πρέπει με την νομοθεσία που θα δημιουργήσουμε να μην ε, δημιουργήσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας ενός σκιώδους τραπεζικού συστήματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι θέλουν να παρέμβουν. Θα ακούσουμε πρώτα τους σκιώδεις εισηγητές της Επιτροπής ΕΚΟΝ και μετά της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και καλό θα ήταν να κρατήσετε το όριο των δύο λεπτών για τις παρεμβάσεις σας έτσι ώστε να μας φτάσει ο χρόνος. Αλλά πιστεύω πως έχουμε αρκετό χρόνο έτσι κι αλλιώς. Κύριε Έγγελ, έχετε πρώτο το λόγο ως και εισηγητής της Επιτροπής. Ευχαριστώ Κίνγκα, ευχαριστώ και στους ε, δύο εισηγητές. Συνεχίζω από αυτά που περιέγραψε η συνάδελφος και φίλη. Η δημιουργία αυτού του Μητρώου στην πραγματικότητα δεν είναι παρά η συνέχεια της πρακτικής που ακολουθείται σήμερα. Δηλαδή, η αρχές που ασχολούνται με αυτό το θέμα με οποιοδήποτε τρόπο, είτε από οικονομική πλευρά είτε από καταπολέμηση του εγκλήματος, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Και αυτό είναι λογικό. Γιατί εν τέλει αυτός είναι ο σκοπός ύπαρξης αυτών των αρχών. Αλλά επιμένω, μιλάμε για αρχές. Δηλαδή για δημόσιες αρχές οι οποίες ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά. Δεν βλέπω κανένα λόγο, κανένα, και κανένα επιχείρημα για το οποίο θα μπορούσε να, με το οποίο θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι κάποιο, οποιοδήποτε άλλο, πέρα από τι αρχέ, θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Επειδή, για παράδειγμα, του φαίνεται ενδιαφέρον και διεξάγει μια δημοσιογραφική έρευνα. Φανταστείτε που θα φτάναμε εάν ε, συνεχίζαμε στην ίδια κατεύθυνση. Για παράδειγμα, οι εισηγμένες εταιρείε στη Γαλλία έχουν την Ε, έχουν με βάση το, το εταιρικό δίκαιο να γνωρίζουν. Φανταστείτε τι θα κάνανε μάλλον εάν, ε, αν είχαν τη δυνατότητα εάν τους ζητούσαμε να μπορούν να ταυτοποιήσουν τους μετόχους τους. Είναι αδύνατο. Τώρα θα μου πείτε ότι είναι λάθος αυτό το σύστημα. Ναι, αλλά υπάρχει. Επομένως δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε εμπόδια και προσκόμματα σε αυτό το, το σύστημα, έτσι κι αλλιώ σίγουρα όχι μέσω μια νομοθεσία η οποία δεν δημιουργήθηκε για να δημιουργήσει προσκόμματα στο σύστημα αυτό. Δεν θα ήταν λογικό. Οι αρμόδιε αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν τον πραγματικό δικαιούχο με τα ε, ε, μέσα που θα τους ε, δώσουμε, που θα έχουν στη διάθεσή τους. Αλλά μόνο εκείνες, κανένας άλλος. Δεν βλέπω επιχειρήματα υπέρ του, της αντίθετης άποψης. Τώρα, μία αναφορά στα λεγόμενα πολίτη στα δημόσια πρόσωπα. Εδώ δεν μιλάμε για άτομα τα οποία συμμετέχουν στην πολιτική. Μιλάμε ε, Ο λόγος για τον οποίο θα θέλαμε να τους ελέγχουμε περισσότερο είναι επειδή θεωρούμε ότι διατρέχουμε περισσότερο τον κίνδυνο διαφθοράς. Στην χώρα μου, συνολικά η οικογένεια θεωρείται δημόσιο πρόσωπο. Δηλαδή όχι μόνο πολιτικός, αλλά και οι ε, συγγενείς του και αυτό δεν το βρίσκω λογικό. Γιατί ο πολιτικός πράγματι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαφθοράς. Μια άλλο παράδειγμα μου σας φέρω, ναι. ο διοικητής ενός δημόσιου οργανισμού, ο διοικητής ενός λιμανιού, αν και δεν έχει πολιτικό ρόλο, μια χαρά θα μπορούσε να συμμετάσχει σε διαφθορά. Και το κείμενο που έχουμε ενώπιον μας δεν το καλύπτει. Δεν καλύπτει αυτή την περίπτωση. Προσωπικά γνωρίζω φίλους μου, δημοτικούς συμβούλους, που αναγκάζονται οι γυναίκες τους να υποβάλουν αναλυτικές δηλώσεις ε, πούμε το βρίσκω λίγο υπερβολικό αυτό. Και τώρα δύο λόγια για την αξιολόγηση κινδύνου. Ναι, είναι απαραίτητη. Αλλά και πάλι υπάρχουν στοιχεία που τα βλέπω υπερβολικά, βρίσκω υπερβολικά για παράδειγμα. Να θεωρούμε ότι οποιοδήποτε τυχερό παιχνίδι στοιχήματα ή online στοιχήματα ή οτιδήποτε τέτοιο. Να θεωρούμε ότι όλα αυτά τα τεχνικά, τυχερά παιχνίδια είναι εργαλεία ξεπλήματος ε, χρήματος και εσόδων από κλιματικέ δραστηριότητες, ούτε αυτό το βρίσκω λογικό. Πρέπει να αξιολογούμε την κάθε κατάσταση κατά περίπτωση για να αναλύσουμε το πραγματικό κίνδυνο που αντιπροσωπεύει. μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα ως το πλαίσιο ε, συγκεκριμένης νομοθεσίας, περιορισμένης στα συγκεκριμένα ζητήματα και όχι ε, να πάμε πιο παραπέρα. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στο σκιώδη συγγετή της ΕΚΟΝ, ο κύριος Σάιμον. Μάλλον ε, στην κυρία Κλίβα η οποία τον ε, αντικαθιστά. Ναι. Ο συνάδελφός μου, ο Πέτερ Σίμων, θα ήθελε να ζητήσει συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ σήμερα. Είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Όμως, καλωσορίζει το σχέδιο της κοινή έκθεση. Θα ήθελε να σε ευχαριστήσει και τους δύο εισηγητές για τη δουλειά τους και με χαρά του βλέπει τις ε, ανησυχίες που είχε ο ίδιος να ε, φαίνονται στο σχέδιο έκθεσης από τους ε, δύο εισηγητές και να έχουν ληφθεί υπόψη στο νέο σχέδιο έκθεσης. Οι ανησυχίε αυτές ήταν ε, η έλλειψη μιας ε, κοινή εκτίμησης κινδύνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και ενός μητρώου επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων και ε, για την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους. Χρειάζεται να βρεθεί ένας κοινός παρανομαστής για, το ξέπλυμα χρήματος. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μία ε, εκτίμηση ε, και μία αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την θέση σε ισχύ της οδηγίας. Έπειτα θα ήθελα να προτείνει όσον αφορά τις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και για την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Και το μητρό αυτό να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τις εισηγμένες του χρηματιστήριο εταιρείε, αλλά όλες τις νομικές οντότητες, ιδρύματα ή διάφορα ή διάφορα τετράστ. Ο κύριος Σίμων θεωρεί πως η πρόταση της Κομισιόν ε, δεν συμπεριλαμβάνει στην πλήρη εκτασή της την εκτίμηση κινδύνου που χρειάζεται και έχει προτείνει μία ε, διαφορετική προσέγγιση, μία απλοποιημένη διαδικασία δέουσας επιμέλειας, ωστόσο Ορισμένα κράτη-μέλη ήδη ενδεχομένως να έχουν ε, αντίστοιχους ε, κανόνες οι οποίοι θα καταστήσουν περί τον ένα τέτοιον κανονισμό, για παράδειγμα σχετικά με τις ε, μεταφορές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς πάνω από ένα ποσό ή ποσά από τυχερά, κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξαιρούνται ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες ή ορισμένοι δικαιούχοι από την διαδικασία της θεούσας επιμέλειας. Αυτό θα διευκολύνει την ε, εκτίμηση του κινδύνου. Ωστόσο, πρέπει να ενημερώνεται σχετικά η ορισμενοι δικαιουχοι απο την διαδικασια της θεουσα επιμελειας αυτο θα διευκολυνει την Επιτροπή για τις εξαιρέσεις αυτές. Και παρά τις προσπάθειές μας ε, για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος, ε, αυτό εξακολουθεί και επιμένει σε μεγάλη κλίμακα. Χρειάζεται επίσης ε, να εξετάσουμε την εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη-μέλη ξεχωριστά και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δούμε ποια βήματα και ποιες ενέργειες έχουν κάνει τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να ε, βοηθήσουν στην επίτευξη του ε, στόχου αυτού της καταπολέμησης ε, του ξεπλήματος χρήματος. Και ο κύριος Σίμων θα υποβάλει τις αντίστοιχες τροπολογίες γραπτός. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρεβάν. Κύριε Μπόσκουιτ, της και γύτρια της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τους δύο εισηγητές για την εξαιρετική τους έκθεση. Το θέμα των μητρώων πράγματι θα αποτελέσει μείζωνα πρόοδο κατάρτιση αυτού του μητρώου που εμείς θέλουμε να είναι δημόσιο βέβαια ή τέλος πάντων να, να έχει πρόσβαση το κοινό. Βέβαια μετά θα δούμε σε ποιο βαθμό θα έχει πρόσβαση το κοινό οι δύο συγγητές μεταξύ τους θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία. Εμείς πάντως θα θέλαμε να είναι ως το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα αυτό. Επίσης, θα θέλαμε ξεκάθαρα να πούμε ότι θα πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ αφενός της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής σφαίρας, κατ' επέκταση, και της καταπολέμησης ε, του ξεπλήματος χρήματος αφετέρου. Στην έκθεση αυτή Καλό είναι που γίνεται λόγος για τους φορείς αυτούς οι οποίοι θα πρέπει να ε, μπορούν να φέρουν τα καθήκοντά τους σε δηλαδή τις ε, μονάδες ε, οικονομικής πληροφόρησης. Επίσης για τους ορισμούς. είναι το φορολογικό αδίκημα σε κάθε χώρα. Πρέπει να βρούμε έναν ορισμό ή τέλο πάντων αν δεν υπάρχει κοινό τόπο μεταξύ των κρατών μελών να καταλήξουμε σε μεγαλύτερη εναρμόνιση. Και τώρα αναφερθώ κάτι σε κάτι που το έχω ξαναπεί. Αυτά τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια. Είναι σημαντικό το θέμα και συμφωνώ να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ιδίως ε, στο θέμα του στοιχηματισμού, γιατί τα παράνομα, ε, μάλλον τα στημένα παιχνίδια είναι ε, ένας τρόπος ξεπλήματος χρήματος. Καλό θα ήταν λοιπόν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο αυτό νομοποίησης στον παράνομες δραστηριότητες. Και ένα τελευταίο. συνεργασία με την ε, Europol, την Ευρωπαϊκή Αστυνομία. Περιλαμβανόταν στην αρχική πρόταση της Κομισιόν και απεσύρθη. Περίεργο φαίνεται αυτό. Γιατί η Europol, όπως και να έχει, συνεργάζεται με τις μονάδες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος. Γιατί λοιπόν αποσύραμε αυτή την αναφορά. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τώρα θα έπρεπε να δώσω το λόγο κανονικά στο σκιώδη εισηγητή Νίλς Τόρβαλτ από την Άλντε που δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος που τον αντικαθιστά. Ουχή. Άρα, κυρία Γκάλ, ούτε το σκιώδη εισηγητή από την Άλντε τον βλέπω. Και δεν υπάρχει μάλλον κανένας που να τον αντικαθιστά ούτε αυτό. Άρα, να δώσω τώρα στον κύριο Γκίγκολτ, την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, που είναι σκιάζει του πρασίνου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα να πω ότι όσον αφορά την οδηγία αυτή, εμείς είμαστε υπέρ ενός δημοσίου μητρώου, ενός ανοιχτού μητρώου και θεωρούμε πως ε, δεν είναι καλή ιδέα αυτό να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Διότι έτσι θα υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα διαφορά συστήματα ελέγχου. Είδατε και πού οδήγησε αυτό στις Ηνωμένε Πολιτείε, όπου τα Μητρό είναι τελείως διαφορετικά. Και μετά οι εταιρείε πηγαίνουν και καταχωρούνται στην Εβάδα ή στο Delaware, όπου τα πρότυπα είναι πολύ λιγότερο αυστηρά. Χρειάζεται να έχουμε ένα κοινό μητρό και είναι φυσιολογικό έτσι κι αλλιώς στην επιχειρηματική ζωή. Όταν ε, ε, επικοινωνείς με μια εταιρεία θέλεις να ξέρεις με ποιον συνομιλείς. Όπως και όταν συνομιλείς με κάποιον ε, άνθρωπο θες να ξέρεις τι είναι αυτός. Τώρα σε περίπτωση ιδρυμάτων δεν έχει ιδέα με ποιον συνομιλείς και πρέπει αυτές οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες. Γι' αυτό πιστεύω πως είναι καλό ότι έχουμε προτείνει έναν τέτοιο διακανονισμό, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός όσον αφορά ε, την, το, τις ε, αρχές ελέγχου. Έπειτα, όσον αφορά το τι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτό το Μητρό, εμείς έχουμε προτείνει ε, τροπολογίες για το θέμα αυτό, αλλά το σημαντικότερο πιστεύω που δεν έχει συζητηθεί ακόμα είναι όσον αφορά την ε, νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματο. Ο στόχο δεν είναι μόνο να βελτιώσουμε τον νόμο, είναι να βελτιώσουμε την εφαρμογή του νόμου. Τώρα, τη Δευτέρα, μόλι, με επισκέφτηκαν ε, αντιπρόσωποι από, τις, ε, από τα αστυνομικά συνδικάτα τη Αυστρία, Γερμανία και τη Ελβετία και μου είπαν ότι υπάρχουν περιπτώσει στι οποίε είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί η νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματο. Δεν αρκεί λοιπόν να κάνουμε πιο αυστηρή νομοθεσία. Έχουμε αρκετή ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρξουν ε, στο μέλλον και να μην επαναληφθούν περιπτώσει όπω αυτέ τη Κύπρου. Πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε η νομοθεσία να επιβάλλεται και να εφαρμόζεται. Και φυσικά υπάρχουν και οι διεθνεί ε, διαδικασίε, όμω και η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα και να διασφαλίσει ότι όπως ακριβώς γίνεται με τα επισητιστικά σκάνδαλα που υπάρχουν διεθνείς έλεγχοι, να φροντίσουμε να επιβάλλονται και να εφαρμόζονται οι νόμοι και να μην είναι απλώς τα χαρτιά, έστω και αν είναι μεταφρασμένα σε 23 γλώσσες. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κέρκ και ο εισηγητής της Επιτροπής ΛΥΠΕ. Ευχαριστώ. Όπως το γνωρίζετε, ε, είμαι εισηγητής για το δεύτερο θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Επομένω, ορισμένε από τι παρατηρήσει μου θα τι αναφέρω σε εκείνο το σημείο. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω κυρίω την κυρία Κεντίνη για το έργο τη από την πλευρά τη ΛΥΜΕ. Η πολιτική μα ομάδα γενικά συμφωνεί και υποστηρίζει την προσέγγιση. Έχουμε του ίδιου στόχου. Μια-δύο παρατηρήσει θέλω να κάνω. Μια και Λείπει ο κύριος Τρέιτσικ, ο οποίος ήταν ο Σχιώδης από την πλευρά της ΙΚΟ και μου έχει ζητήσει να μεταφέρω και κάποια στις του παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, τα δημόσια πρόσωπα. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος προσωπικά αισθάνομαι λιγάκι άβολα ως δημόσιο πρόσωπο. Υποστηρίζουμε το γεγονό ότι χρειάζεται η ε, εξεργασία προσωπικών δεδομένων για να εντοπίζονται ποια είναι αυτά τα, τα δημόσια πρόσωπα, αλλά δεν συμφωνούμε να συμπεριλαμβάνεται η οικογένειά τους θα πρέπει να περιοριζόμαστε στις ε, ατομικές και επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι διεφθαρμένα δημόσια πρόσωπα προφανώς ε, θα πρέπει να ταυτοποιούνται και θα πρέπει να ταυτοποιούνται και από τις εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν την ανάλυση ρίσκου, αλλά αυτό δεν συμπεριλαμβάνει τα μέλη των οικογένειών τους. Τώρα, σχέση με τον πραγματικό δικαιούχο, αναφέρεται ότι θα πρέπει να παρέχονται αυτά τις πληροφορίες μέσα σε 30 ημέρες, αλλά θα χρειάζεται μια ευελιξία αυτό, γιατί ορισμένες φορές χρειάζεται να περιμένουμε τις πληροφορίες που οι εταιρείε υποβάλλουν κάθε, σε ετήσια βάση και αυτές οι πληροφορίες ίσως μας δώσουν μεγαλύτερη ακρίβεια. Τώρα, σε σχέση με τη φοροδιαφυγή, Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και τους φορολογικούς παραδείσους, όπως επίσης και την, ε, ε, μαζί με την καταπολέμηση του ξεπλήματος. Δεν υπάρχει καμία αντίθεση, αντιθέτως αυτές οι δύο δραστηριότητε είναι συμπληρωματικέ. Τώρα όσον αφορά την κοινοποίηση και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων πριν ε, συλλεγούν στοιχεία που τους αφορούν, θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο αυτή η ενημέρωση πιθανόν θα υπονομεύσει τη διαδικασία. Τώρα, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν, να δίνουν ένα feedback για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν αυτά τα στοιχεία που τους παρέδωσαν εταιρείε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουν αναδείξει και πολλές εταιρείε. Το θέμα τώρα της προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι όποιες ρυθμίσεις θα πρέπει να βασίζονται σε μια ανάγκληση ρίσκου και να είναι πρακτικά εφαρμόσιμες. για να είναι αποτελεσματική αυτή η λύση θα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί και να μην δημιουργεί προβλήματα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή στους ιδιώτες οι οποίοι απλώς θέλουν να ανοίξουν έναν λογαριασμό. Ο στόχος μας πρέπει να ε, συλλάβουμε τους εγκληματίες ε, που είναι ε, υπόλογοι για σοβαρά δικήματα, όχι να δυσκολέψουμε τη ζωή κάθε πολίτη. Να μην κάνουμε τα ίδια λάθη που έχουμε κάνει με προηγούμενες οδηγίες σε σχέση με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και δυσκόλεψε τη ζωή πάρα πολλών καταναλωτών. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο το ξεχνούμε. Αλλά επίσης, κατά την άποψή μου, θα πρέπει ταυτόχρονα να σκεφτόμαστε τους πολίτες οι οποίοι κατά τεκμήριο τηρούν τον νόμο και δεν θα πρέπει να τους ταλαιπωρούμε χωρίς λόγο και αιτία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σκιώδης εισηγητής για την ΚΟΕ, κ. Κλουτ. Δεν είναι εδώ, μήπως τον αντικαθιστά κάποιος. Όχι. Κυρία Γκάρλα, ποιον έχετε εσείς ως εκπρόσωπο της ΚΟΕ. Δεν είναι εδώ εκπρόσωπος της ΚΟΕ την πλευρά της ΕΚΟΝ. Όχι. Ε, κλείσαμε λοιπόν με τους σχεδόν συζητητές και δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Μάρτιν Φρούν, ils ont mal noté cela. Συγγνώμη, δεν ε, ήξερα ακριβώ ποιο είναι το όνομά σα. Είστε εδώ, είμαι εδώ. Δεν υπάρχει και πρόβλημα και με το όνομά μου, κυρία Πρόεδρε. Κατάλαβα ότι πρόκειται για μένα. Θα τα πούμε στα αγγλικά. Και γιατί πιο πολλές παρεμβάσεις έγιναν στα αγγλικά, γιατί αυτήν την γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Καταρχάς, ε, θερμές ευχαριστίες ε, στους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές. Καλή, ενδιαφέρουσα και ενθαρρυντική η έκθεση που είμαι βέβαιος θα βελτιωθεί ακόμη περαιτέρω όσο θα προχωρούν οι εργασίες της Επιτροπής σας ή των Επιτροπών σας καλύτερα. Νομίζω ότι αυτά τα τέσσερα ζητήματα που ανέφεραν οι κύριοι Κάρεν Σαρτζεντίνη είναι και τα πλέον ε, σημαντικά της ε, πρότασής μας. Εν συντομία θα ήθελα να αναφερθώ και στις εξελίξεις σε αυτό το τομέα για τις εργασίες δηλαδή που εμείς ε, αναλαμβάνουμε και με την Προεδρία και με τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά το Μητρό των Πραγματικών Δικαιούχων, πολύ δραστηριότητα και στην G8 και στην G20 με επικεφαλή στο Ηνωμένο Βασίλειο που προείσταται και των εργασιών του Συμβουλίου στο θέμα αυτό. Ε, πιστεύω ότι υπάρχει έτσι μια κίνηση. Να ξεκαθαρίσω ότι εμείς δεν είχαμε προτείνει κάτι τέτοιο, είχαμε προτείνει ένα πρώτο βήμα ότι θα μπορούσε να υπάρξει υποχρέωση για τις επιχειρήσεις σε περίπτωση που χρειαζόταν να αποκαλυφθούν κάποια στοιχεία. Όταν δηλαδή ιδίω η επιχείρηση έχει κάποια πολύπλοκη δομή να δίνονται πληροφορίες. Εμείς δεν λέγαμε ότι θα πρέπει κάθε εταιρεία που έχει πολύπλοκη δομή και διαστρωματώσεις να έχει αυτό το μητρό. Αλλά πάντων εμείς είχαμε προτείνει το πρώτο βήμα. Δεν είχαμε φτάσει στο σημείο του δεύτερου, της πρώτης αυτής στο δεύτερο βήμα. Δηλαδή θέλαμε εμείς να υπάρχει αυτή η υποχρέωση και μετά τα κράτη-μέλη θα αποφάσιζαν πού θα συλλέγονται αυτές τις πληροφορίες. Εμείς είμαστε ανοιχτοί να βελτιώσουμε το κείμενο και να περάσουμε σε υποχρέωση των κρατών μελών να δημιουργήσουν ένα είδος ε, μηχανισμού κεντρική αποθήκευση και εύκολη πρόσβαση ε, στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων. Είναι μεγάλη συζήτηση βέβαια και στις δηλώσεις Νομίζω το αναφέρατε και εσεί, δηλαδή είναι μεγάλη συζήτηση του κατά πόσο οι υπερφορέ αυτέ θα πρέπει να είναι δημόσιε και θα μα ενδιαφέρει πολύ να δούμε προ τα που ε, θα βαδίσετε. Είμαστε ανοιχτοί πάντω. Να πω κάτι που δεν αναφέρθηκε, άρα θα έπρεπε να αναφερθεί, σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων. Όταν μιλάμε για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν δημοσιεύονται στοιχεία για ε, τα, τα, τα περιουσιακά στοιχεία κάποιου. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ υπάρχουν αξιολογότατοι βουλευτές που τα γνωρίζουν τα πράγματα πολύ καλά. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα θέμα λίγο λεπτό. Για αυτά τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα. Είναι αρκετά ευρύ το παιδί ε, και το εύρος φτάνουμε μέχρι το τοπικό επίπεδο ουσιαστικά. Μπορεί να μην αφορά βέβαια τον κάθε τοπικό σύμβουλο, αλλά αφορά σίγουρα τους δημάρχους. Ο δήμαρχος θα μπορούσε να αποτελέσει ε, πιθανό, ενδεχό, πιθανό θύμα ε, δωροδοκίας. Αυτά τα στοιχεία για αυτά τα άτομα θα πρέπει να επικαιροποιούνται. Υπάρχουν ε, και πολύ, σε τοπικό επίπεδο, πολλά το, έτσι, δημόσια, πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, όπως τα λέμε στην πρότασή μας. Ίσως χρειαστεί δηλαδή ένταση πόρων για τη συγκέντρωση όλων αυτών των στοιχείων σε επίπεδο κράτους μόλις πόσο μάλλον σε επίπεδο κομισιών. Γι' αυτό λοιπόν κάπως ε, πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε με αυτή την ιδέα που επαναλαμβάνω απαιτεί και ένταση πόρων, μια ευρωπαϊκή λίστα πολιτικών προσώπων, που πρέπει να επικαιροποιείται συνεχώς όπως είπα. Αξιολόγηση κινδύνων. Και εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη μας μια εξέλιξη και από πλευρά κρατών μελών, δηλαδή ότι ζητείται ε, ανάληψη δράσης και συμμετοχή από την Κομισιόν. Υπάρχουν τα όρια που ε, μας διέπουν και σίγουρα πρέπει να έχουμε συντονισμό και με τα κράτη-μέλη. Γιατί υπάρχουν εμπειρογνώμονες ε, που γνωρίζουν επιτόπου καλύτερα ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Θα πρέπει να δούμε πώς οργανώσουμε την όλη διαδικασία. Σε αυτή τη φάση θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσέξετε λίγο το θέμα του χρονοδιαγράμματος, ε, του timing. Η εξολόγηση των κινδύνων δεν είναι κάτι εύκολο ως εγχείρημα. Σε κάποιες χώρες ήδη έχει ξεκινήσει σχετική δουλειά, αλλά σε κάποιες άλλες καθόλου. Η Κομισιόν επίσης δεν έχει ίσως την απαιτούμενη εμπειρία και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε επαρκή χρόνο στη διάθεσή μας για να ε, φέρουμε σωστά σε πέρα σε αυτό το εγχείρημα. Υπάρχουν θέματα που αφορούν άμεσα την ε, νέα αγορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε δύο χρόνια που είναι περίοδος εφαρμογής και εκεί πρέπει να γίνουν αξιολογήσεις κινδύνων. Μια ρεαλιστική προθεσμία, ένας χρόνος νομίζω ότι είναι λίγο. Δεν είναι σχεδόν τίποτα δηλαδή αν λάβει υπόψη κανείς πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Προστασία δεδομένων. Μας ικανοποιεί το ότι όλη οι αξιολόγηση έκανε και την Κομισιόν να προτείνει όχι ένα ειδικό καθεστώς προστασίας δεδομένων, αλλά κάτι που να συνδέεται με την υφιστάμενη νομοθεσία. Συμφωνούμε, ε, μάλλον ε, χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι και οι συνεισηγητές προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Με να δούμε περιπτώσεις, συνθήκες, περιστάσεις όπου μπορούμε να είμαστε ίσως πιο συγκεκριμένοι, να προσθέσουμε μεγαλύτερη σαφήνεια. Ας συνεργαστούμε λοιπόν με τους εισηγητές και άλλους βουλευτές για την περαιτέρω βελτίωση του τμήματος αυτού της πρότασής μας. Διατρέχω τις σημειώσεις μου για να δω αν θα έπρεπε να σας σχολιάσω κάτι ακόμη. Ακούστηκε κάτι για εξαιρέσεις για κάποιους παρόχους, για κάποιες δραστηριότητες. δεν ε, θέλουμε να υπάρχουν σαφείς παρεκκλήσεις. Ε, δεν είναι τουλάχιστον ε, κάτι που προβλέπεται στα διεθνή πρότυπα που εμείς θέλουμε να τηρήσουμε. Θέλουμε να έχουμε αυτή την προσέγγιση βάσει των κινδύνων, risk-based approach, αλλά όχι να έχουμε πολύ σαφείς εξαιρέσεις ή παρεκκλήσεις θέλαμε να είναι σε πάρα πολύ εξαιρετικέ περιπτώσεις. Για κάποιες δραστηριότητες, ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ανοιχτοί προς πλήρη εξαίρεση ή έστω μερική εξαίρεση. Θα δούμε ποιοι τομείς θα μπορούσαν να είναι αυτοί και θα συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Επίσης παρατήρηση για τους ε, πόρους, ε, για τις μονάδες αυτές της χρηματοοικονομικής προφόρησης συμφωνούμε. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τη Europol, αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει συζήτηση. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με την νομική βάση της οδηγίας αυτής όταν ε, πραγματευόμαστε ζητήματα που αφορούν την συνεργασία σε ποινικά θέματα. Γι' αυτό και είδαμε λίγο κριτικά της περίληψη της αναφορά στην Europol. Πρέπει να δούμε την νομιμότητα, δηλαδή την νομική βάση. Εκεί υπάρχει ως ένα πρόβλημα. Επίσης, συμφωνώ πολύ με αυτό που είπε ο κύριος Κέρκοπ, να είμαστε ανάλογοι, να μην είμαστε δυσανάλογοι μάλλον και να μην επιβάλλουμε πολύ μεγάλο βάρος σε επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να είναι αναλογικός ο τρόπος εφαρμογής στους υποχρέους, στις υποχρέες οντότητες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αν θέλετε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την πρόταση. Πέρασα κατά πολύ τα πέντε λεπτά, αλλά τέλος πάντων ε, έπρεπε να τα πω όλα αυτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ποιο άλλο ε, βουλευτή θέλει να λάβει το λόγο. Έχω στον κατάλογο μίδι την κυρία Γκόμε. Κυρία Λούλινγκ θέλει επίση το λόγο. Λοιπόν, κυρία Γκόμες, πρώτα και μετά κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Συνεργάζομαι με την Πορτογαλική Εισαγγελία για να αποκαλύψω ένα σκάνδαλο διαφθοράς όσον αφορά την πώληση κάποιων γερμανικών υποβρυχίων στην Πορτογαλία. Καταρχάς, ε, πρέπει να δούμε τις τράπεζες που ήταν ε, αναμεμειγμένες στην όλη ιστορία και κοιτάζοντας όλον αυτόν τον ιστό καταλήγω και εγώ, όπως και όλοι οι συμπολίτε μου, ότι το σύστημα είναι σχεδιασμένο, ειδικά για τη διαφθορά. Είναι σχεδιασμένο για να ξεπλύνεται χρήμα. Γι' αυτό είναι απολύτω απαραίτητη μια τέτοια οδηγία. Και συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους που είπαν ότι, με τον κύριο Γκίγκολ μάλιστα, που είπε ότι χρειάζεται ένα ε, δημόσιο, ανοιχτό, προσβάσιμο μητρό καταχώρηση. Διότι σας είπα, το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να χρησιμοποιείται για ε, απόκρυψη χρημάτων, για διαφθορά, για ξέπλυμα και για φοροδιαφυγή. Όσον αφορά τώρα τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, ναι. Και εγώ υπήρξα δημοτική σύμβουλος και φυσικά και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και δημοτικοί σύμβουλοι στα Μητρώα αυτά. Έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες ε, διαφθοράς. Δεν πρέπει να ξεφεύγει κανένας από αυτό το μητρό. Πρέπει επίσης να λαμβάνουμε υπόψη ότι οι εποπτικές αρχές, όπως για παράδειγμα οι κεντρικές τράπεζες, δεν επιτρέπεται να απασχολούν ε, άτομα με τα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, όπως γίνεται στην Πορτογαλία, στη χώρα μου. Επίσης, θα νόμιζε κανείς ότι τα πράγματα στην Πορτογαλία είναι πολύ καλύτερα από ότι εκτός. Όμω ξέρετε πώς μα λένε στην Αγκόλα, πλυντήριο. Η χώρα μου χρησιμοποιείται για να ξεπλένατε χρήμα. Και μην ξεχνάτε ότι η χώρα μου επίσης είναι μια χώρα όπου από τις 20 εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείε οι 19 δεν έχουν κάποια μητρική εταιρεία με έδρα στην Πορτογαλία. Κάποιες είναι στις νήσους Καϊμάν, κάποιες στην ε, Ελβετία. Μόνο μία έχει την έδρα της στην Πορτογαλία και δεν τρέπονται καθόλου γι' αυτό. Διότι έχουν τα κεντρικά τους ε, σε κάποιες, ε, ακόμα και ευρωπαϊκές χώρες όπως οι για παράδειγμα, η Ολλανδία, όχι μόνο πληρώνουν λιγότερους φόρους, αλλά και μπορούν πάρα πολύ εύκολα να κρύψουν τα κέρδη που αποκτούν στην Αγκόλα, στη Βραζιλία, στη Μοζαβίκη, όπου τα αποκτούν. Και φυσικά αυτό δεν είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Πορτογαλίας, όλοι το κάνουν. Δεν, μην περιμένετε λοιπόν να καταπολεμήσουμε την εφοροδιαφυγή και την διαφθορά με έτσι, απλές οδηγίες. Έγινε μια συμφωνία με την Ελβετία και να σας πω κιόλας ότι βρέθηκαν πάνω από 4 δισεκατομμύρια στην Ελβετία που ανήκαν σε πορτογαλικές εταιρείες. Τους δόθηκε λοιπόν αμνηστία παρότι αποκαλύφθηκαν αυτές οι παρανομίες και όχι μόνο έπρεπε, χρειάστηκε να πληρώσουν λιγότερο φόρο από αυτόν που έπρεπε να πληρώσουν, αλλά δεν χρειάστηκε ούτε καν, δεν τους υποχρέωσαν να επιστρέψουν τα χρήματα που είχαν καταχωνιάσει στην Ελβετία. Και αυτό γίνεται επί εποχή Τρόικας. Γι' αυτό λοιπόν ρωτώ, τι κάνει η Κομισιόν. Γιατί υπάρχουν και μέλη σας στην Τρόικα. Τι γίνεται λοιπόν βασισμένο στην οδηγία, τι γίνεται στα χαρτιά στην οδηγία και τι γίνεται στην πράξη, στην εφαρμογή όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τέλος, να πω ότι δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει η πιο αυστηρή νομοθεσία. Χρειάζεται είναι απαραίτητη η συνεργασία με την Ευρωπόλ. Χρειαζόμαστε εγγυήσεις ότι θα έχουμε εποπτικέ, θα, θα έχουμε αρχές οι οποίες θα είναι ικανές και θα βρίσκονται πριν τους εγκληματίες και όχι από πίσω τους, δεν θα τους ακολουθούν. Πρέπει επίσης να έχουμε δικαστές και εισαγγελείς εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αδιάφθορους και να σας υπενθυμίσω αυτό που είπα πριν για τα γερμανικά υποβρύχια και την πώλησή του στην Πορτογαλία. Να σας πω ότι βρέθηκαν ε, τα σχετικά έγγραφα για αυτές τις ε, συναλλαγές στη Γερμανία και κατασχέθηκαν εκεί. Η κυρία Λούλιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. συχνά παρεμβαίνω στα ζητήματα αυτά. Το ίδιο θα κάνω και τώρα, έχοντας ακούσει τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Πια Ήταν μια από τις σπάνιες φορές που κατάλαβα ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής ήταν πιο λογική από αυτή που έχουμε τώρα επιτάπητος και συμφωνώ πλήρως με αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, κυρίως όσον αφορά την αναλλαγικότητα και την ανάγκη να είμαστε προσεκτικοί. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την κυρία Αργεντίνη στο θέμα του Μητρώου και είπατε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τον πολίτη και ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να πληροφορείται, να γνωρίζει τα πάντα, το ίδιο εσύ για τους δημοσιογράφους, για τους ΜΚΟ. Ναι, εγώ ίδια, ως πολίτης, για ένα παρήργο λόγο δεν αισθάνομαι προστατευμένη. Όταν μου λένε ότι θα υπάρχει ένα μετρό, μέσω του οποίου όλοι θα μπορούν να γνωρίζουν τα περιουσιακά μου στοιχεία. Και αυτό θα, σε αυτό θα έχουν πρόσβαση δημοσιογράφοι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, όποιος θέλει. Κατάλαβα πολύ καλά ότι θέλουμε να αποτρέψουμε την πώληση αυτών των στοιχείων. Αν ακολουθήσουμε όμως την πρότασή σας για, για το Μητρό, ναι, κανείς δεν θα τα πουλάει αυτά τα στοιχεία γιατί όλοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά. Είναι και αυτό μια λύση. Μιλάμε λοιπόν για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του πολίτη. Και θεωρώ ότι το Μητρό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και να έχουν πρόσβαση σε αυτό μόνο οι αρχές. Διαφορετικά τι θα κάνουμε, θα μπορεί ο γείτονά μου να μαθαίνει ακριβώς ποια είναι τα περιουσιακά μου στοιχεία, τι αγόρασε χτες. Νομίζω ότι το παρατραβάμε. Και ιδίω οι πράσινοι, οι οποίοι πάντα είναι στην πρώτη γραμμή όταν μιλάμε για την προστασία του πολίτη και των δικαιωμάτων Τώρα θέλουν όλα στο φως να βρίσκονται. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι απαραίτητο. Ας παραμείνουμε σε ένα πλαίσιο ε, σεβασμού της αναλογικότητας στο θέμα αυτό. Είμαι βέβαιη πάντως ότι οι εισηγητές θα απαντήσουν σε όλα αυτά. Ευχαριστούμε κύριε Αλάλη. Δίνω και πάλι το λόγο στους ε, δύο συνεισηγητές. Αλλά αυτή τη φορά να τηρήσουμε, σας παρακαλώ πολύ, το χρόνο κυρία Κάρινς. Κύριε Κάρινς, πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνάδελφου για τα σχόλιά τους και περιμένω με υπομονησία να λάβω τις τροπολογίες που θα συνοψίζουν ε, με εύληπτο ε, νομικό τρόπο όλα τα επιχείρηματα που ακούσαμε σήμερα. Σε ό,τι αφορά τα φορολογικά εγκλήματα ορισμός. Αν κάποιος θεωρεί ότι ε, χρειαζόμαστε έναν καλύτερο ορισμό, ε, με τα χαράς να δω έναν τέτοιο καλύτερο ορισμό. Είμαι ανοιχτός. Δεύτερον, Europol, η αναφορά στο άρθρο 54 ετέθε ένα θέμα ε, νομικής αιτιολογίας. Δεν το έχουμε έτσι γιατί μας ήρθε ε, διαγράψει, υπήρχε νομική αιτιολογία. Αλλά ναι, να το ξαναδούμε αν θεωρείτε. Για τα τέσσερα τώρα ζητήματα, τους πραγματικούς δικαιούχους, ε, πολιτικώς εκτεθειμένα, πρόσωπα εξόλωσης κινδύνου, προσωπικά δεδομένα. Το βασικό είναι ε, η πραγματική δικαιουχή, το μητρό αυτό. Φαίνεται ότι συμφωνείτε όλοι, αλλά ε, το πρόβλημα που διαβλέπω είναι ότι δεν υπάρχει συμφωνία σε ό,τι αφορά το βαθμό του ανοίγματο. Υπάρχει ζήτημα προστασίας δεδομένων και της ιδιωτικότητας, προστασία της ιδιωτικότητας. Αυτό το θέμα νομίζω θα πρέπει όλοι να το δούμε, όχι συναισθηματικά, αλλά να δούμε τι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις θα έχει. Δεν θέλουμε επενδύσεις και νέες θέσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτοί που έχουν χρήματα για να επενδύσουν έχουν και την επιλογή του πού να επενδύσουν τα χρήματά τους. Μπορούν λοιπόν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση και θέσει εργασίας ή να αγοράσουν ε, μετοχές μιας μεγάλης ε, εταιρεία στο χρηματιστήριο, από τη Siemens και δεν ξέρω εγώ ποια άλλη αμερικανική εταιρεία. Ε, τρίτη επιλογή να αγοράσουν χρυσό ή άλλα διαρκή αγαθά και να τα αποθηκεύσουν σε κάποιες ε, αδασμολόγητες αποθήκες και να περιμένουν εκεί να βγατήσουν. Αν θέλουμε μάλλον με αυτό που λέμε, τους λέμε ουσιαστικά πάρτε τα χρήματά σας και μην τα επενδύσετε σε επιχειρήσεις ε, στην Ευρώπη, πηγαίνετε, τα βάλτε, τα, πηγαίνετε τα κάπου αλλού. Εμείς θέλουμε να σταματήσουμε το ξέπλυμα χρήματος και θα έχουμε ένα τεράστιο δίχτυ για να πιάσουμε ε, τα μεσαία ψάρια, ε, εκατοντάδες χιλιάδες ε, ανθρώπους που θα εκτεθούν και στον τύπο και στους υπόλοιπους. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Αν πετάξουμε ένα τέτοιο, αν ρίξουμε ένα τέτοιο δίχτυ, θα πιάσουμε όχι μόνο τα μεγάλα ψάρια, αλλά και αυτά που δεν θέλαμε να πιάσουμε. Άρα το σκεφτούμε δύο και τρεις φορές πριν καταλήξουμε πάνω σε αυτήν την πρόταση. Θα έχουμε και άλλες συζητήσει σίγουρα με τους σκιώδεις εισηγητές και θα εξετάσουμε και όλες τις τροπολογίες που θα κατατεθούν. Ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ κύριε Κάνης. Κυρία Σαρζεντίνη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η συνάδελφος Μπόσκουρτ δεν είναι εδώ στην αίθουσα, αλλά σε ό,τι αφορά τον ορισμό ε, φορολογικού εγκλήματος ε, ή φορολογικής παράβασης. Δυστυχώς ο ορισμός δεν υπάρχει για το φορολογικό αδικήμα θα χρειαζόταν μια εντελώς διαφορετική βάση. Η χρηματοπιστωτική, η τραπεζική φορή ουσιαστικά εξαρτώνται από την εθνική νομοθεσία για το τι είναι φορολογικό αδίκημα. Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών θα ήταν μια λύση για την καταπολέμηση φορολογικών εγκλημάτων. Βέβαια χρειάζονται άλλες προτάσεις νόμου για κάτι τέτοιο. Αν έχουμε ένα ανοιχτό μητρό ε, των πραγματικών δικαιούχων, κάτι που συζητάμε συνεχώς. Αυτό είναι ένας τρόπος καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Εγώ αυτό ζητώ. Ένα ανοιχτό, ε, ένα δημόσιο αρχείο, μητρό μάλλον. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπόλη, γιατί αποσύρθηκε η πρόταση αυτή. Ακούστε, ο ρόλος της Europol στη διατύπωση η αξιολόγηση των κινδύνων ε, υπάρχει, αλλά εμείς νομίζουμε ότι έγινε συζήτηση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθερών για την εντολή. Δεν μπορεί ένα καζίνο, για παράδειγμα, να δίνει στην Ευρωπόλ στοιχεία για άτομα ε, των οποίων δεν έχει ξεκινήσει κάποια έρευνα μπορεί να δημιουργηθεί μια μονάδα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Μία ασχολείται με το ποινικό δίκαιο, με το αστικό δυνάμει του δικαίου. Αυτές οι μονάδες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης μπορεί να εξαρτώνται ή να συναρτώνται στο αστικό ή στο ποινικό αν όμω δίνει πληροφορίε μια τέτοια μονάδα στις δυνάμεις του νόμου, στι δικαστικέ αρχέ. είναι μια λύση και γι' αυτό δεν αναφερόμαστε στη Europol, σε ό,τι αφορά τον κατάλογο πολιτικώ εκτεθειμένων προσώπων. Γι' αυτό χρειάζεται σίγουρα, χρειάζονται πόροι σημαντικοί και το καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει να βρούμε μια λύση όμω. Για να μην εξαρτώμαστε πια από εμπορικέ εταιρείε. Πρέπει να απεξαρτηθούμε από αυτές τις εταιρείες. τα Μητρώα και οι κατάλληλοι πολιτικώ εκτεθειμένων προσώπων είναι τελείω διαφορετικά μεταξύ του. Μην τα αφομοιώνουμε το ένα με το άλλο, είναι διαφορετικά θέματα. Λούλινγκ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το θέμα για τη συζήτηση για το θέμα αυτό και θα περάσουμε σε ένα άλλο σχέδιο έκθεσης πρόταση κανονισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές ε, ποσών, τα εμβάσματα. Κλέβα και Κύρκοπ δύο συγγητές. Δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Κλέβα καταρχάς. After presentation of... Μετά την παρουσίαση της οδηγίας, θα ήθελα να πω και δύο λόγια για το μικρό αδερφό της οδηγίας αυτής, την οδηγία της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Στην κοινή μας έκθεση ε, μπορώ να πω ότι ΕΚΟΝ, θα, θα μιλήσω μάλλον για τα όσα μπήκουν στην αρμοδιότητα της ΕΚΟΝ περισσότερο και ο συνάδελφος για ε, τα θέματα που μπήκουν στην αρμοδιότητα της ΕΛΥΠΕ. Λοιπόν, είναι ένα διπλό πακέτο, οδηγία και κανονισμός και στα δύο πρέπει να ενισχυθεί η διαφάνεια, ε, η διασυνοριακή και η εθνική, έτσι ώστε να, οι αρχές επιβολής νόμου να μπορούν να εντοπίσουν τι ε, ροές ε, χρημάτων. Η πρόταση κανονισμού, πως και στην οδηγία, προσπαθεί να ακολουθήσει τα διεθνή πρότυπα. Οι προτάσει της Ευρωπαϊκή Επιτροπής σκοπεύουν να διευκολύνουν ε, από τη μία τις ε, μεταφορές ποσόν και από την άλλη να διασφαλίσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμορφώνεται πλήρως με το ΦΑΤΕΦ και με τα διεθνή πρότυπα. Δεν πιστεύω ότι η επικαιροποίηση του κανονισμού από την, από την Κομισιόν ε, είναι, τηρεί μάλλον τη δέσμευση της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα. Στην αναθεώρηση αυτή και οι πληροφορίες για αυτόν που πληρώνει και για εκείνον που δέχεται την πληρωμή ε, απαιτούνται. Πιστεύω πως αυτό αυτό, ε, αυτή είναι η, καλή, η σωστή προσέγγιση έτσι ώστε να ε, διασφαλίζεται ότι θα λαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες. Έπειτα, η προσέγγιση με βάση την εκτίμηση κινδύνου. Είμαι υπέρ αυτή. είναι σημαντικό όμως να ε, δούμε τα επιμέρους σημεία πίσω από αυτή και χαίρομαι πολύ που θα συζητηθεί η ευρωπαϊκή διάσταση ε, της ε, προσέγγισης αυτή και που έχει ληφθεί υπόψη της τόσο από την Κομισιόν όσο και από το Συμβούλιο και εδώ. Όμως ε, δεν γίνεται να έχουμε ελλειπείς πληροφορίες ως τη μόνη βάση, βάσιμη υποψία. Χρειάζεται λοιπόν μια προσέγγιση βασισμένη στις εκτιμήσεις κινδύνου. Οι τράπεζες πρέπει είναι και αυτές σε θέση να εντοπίσουν τις ύποπτες συναλλαγές και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα αυτό ισχύει και για τις ε, μεταφορές ποσών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, εντός ενιαία ενιαίας αγοράς. Έπειτα, διευκρινήσεις σχετικά με τον ε, ρόλο των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών πιστεύω πως η διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που όντως παρέχουν υπηρεσίες και στους ε, διαμεσολαβητές είναι υπαρκτές και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Γι' αυτό με την ε, κοινή μας ε, έκθεση αναφέρουμε ότι ο Μεσάζοντα θα είναι υπεύθυνο για τι ανεπαρκεί ελλειπεί πληροφορίε και θα υπάρχει και ένα σχέδιο Β σε περίπτωση που συμβαίνει αυτό. Ο... Οι υποχρεώσει ε, του όμω πρέπει να είναι ίδιε ε, με τι υποχρεώσει που έχουν και οι τράπεζε από τι οποίε ε, αρχίζει αυτή η μεταφορά των ποσών. Πιστεύουμε επίσης πως η αύξηση των κυρώσεων και πιο αυστηρές κυρώσεις είναι ένα σωστό βήμα ιδιαίτερα για τους παρόχους υπηρεσιών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο εκθέσεις πιστεύουμε ότι βελτιώνουν τους εφιστάμενους κανονισμούς και οδηγίες, αλλά πρέπει όπως και στην προηγούμενη περίπτωση να κοιτάξουν την πραγματικότητα και να υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές που θα διερευνούν παραβιάσεις που έχουν συμβεί εκτός της επικράτειας της Ένωσης. για παράδειγμα, έχουμε και την οδηγία της κεφαλαιακής απαιτήσει 4, έχουμε την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή που θα μπορούσε να ε, επιβάλλει κυρώσεις και κυρώσεις για, ε, σε περιπτώσεις ξεπλήματος χρήματος. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι να δούμε τι, τις ζημιές που ενδεχομένως προκύψουν σε περίπτωση κακής χρήσης του τραπεζικού συστήματο για χρηματοδότηση τρομοκρατία ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε ενέργειες. Πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε και όχι να δημιουργήσουμε παρετέρω εμπόδια στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Γι' αυτό λοιπόν σα ε, ε, εφιστώ την προσοχή σε αυτό. Ε, τέλος, θέλω ήθελα να ευχαριστήσω τον συνεισηγητή μου, κύριο Κέρκοπ, για την καλή συνεργασία και ε, χαίρομαι για την μελλοντική μας συνεργασία και για τις τροπολογίες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κλέβα. Ο κύριος Κέρκοπ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ε, θα προσπαθήσω να μην επαναληφθώ, γιατί Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με όσα είπε η συναδελφός μου και συνεργαζόμαστε εξάλλου στενά. Θα ήθελα να τονίσω κάποια σημεία από τη σκοπιά της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, διότι κατά την άποψή μου και έτσι κι αλλιώς έχω ασχοληθεί πολύ με νομοθετικού περιεχομένου ζητήματα στην καριέρα μου για την καταπολέμηση της, του ξεπλήματος χρήματος και στο Ευρωκοινοβούλιο και ως υπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο στο παρελθόν. Πιστεύω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εφαρμογή νομοθεσίας. Γι' αυτό, όπως είπα και νωρίτερα, η προσέγγιση μας θα πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε έναν ε, αναλογικό ε, και κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης της, ε, του ξεπνήματος χρήματος και να μην δημιουργήσουμε πρόσθετα εμπόδια. Γι' αυτό και στηρίζω απόλυτα την προσέγγιση βασισμένη στην εκτίμηση κινδύνου όπως ανέφερε και η κυρία Σαρτζεντίνη λίγο πριν, μια τέτοια προσέγγιση βοηθά διότι εξετάζει τους κινδύνους σε κάθε τομέα. Και το τονίζω αυτό γιατί υπάρχουν ε, ορισμένοι τομείς οι οποίοι ε, είναι πολύ χαμηλού κινδύνου και πιστεύω πως αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη στις προτάσεις μας. Επίσης, καλωσορίζω την ε, δυνατότητα δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Το οργανωμένο έγκλημα κοστίζει στον Ευρωπαίο φορολογούμενο δισεκατομμύρια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε λογικοί, συνετοί και να χρησιμοποιήσουμε τους υφιστάμενους κανόνες. Το ξέπλυμα χρήματος είναι μία από τις ε, χειρότερες παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδοτεί ορισμένα από τα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα, συμμορίες, εμπόριο όπλων, διακίνηση ανθρώπων. Πρέπει λοιπόν να κλείσουμε τις ε, κάνουλες από τις οποίες ρέει το χρήμα προς αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις. Και ε, η δυνατότητα κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων θα μειώσει την ε, δυνατότητα χρηματοδότησης των ε, εγκληματικών αυτών οργανώσεων και πιστεύω ότι οι φυστάμενες και ελπίζω μελλοντικέ συμφωνίες ε, εμπορίου και επενδύσεων θα συμπεριλαμβάνουν τέτοιες διατάξεις και θα βοηθήσουν την Ευρώπη να αναπτυχθεί, να ευημερήσει αλλά και να καταπολεμήσει το έγκλημα και αναφέρομαι στο χρηματοπιστωτικό έγκλημα δεν θα επεκταθώ στο κυβερνό έγκλημα διότι δεν χρειάζεται να να σας πω εγώ πόσο πολύ κοστίζει και θα συνεχίσει να κοστίζει όλο και περισσότερο το κυβερνό έγκλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως επιτοπλίστων αρκετά καλή νομοθεσία. Γιατί λοιπόν δεν εφαρμόζεται σωστά. Πιστεύω πως με το να εναρμονίσουμε τον ε, κανονισμό αυτό με τους ε, κανόνες FTTF, ε, με την οδηγία για τις τραπεζικές πληρωμές, είναι... θα μπορέσουμε να κάνουμε το σύστημα πιο αποτελεσματικό. Φυσικά, χρειάζεται επαλήθευση του ονόματος των, των, των συναλλαγών για συναλλαγές πάνω από 1000 ευρώ. να λάβουμε υπόψη το άρθρο 8 και να ε, φροντίσουμε για την καλή συνεργασία μεταξύ των αρχών που αναφέρεται στο άρθρο 22. Επίσης να πω ότι οι υπερβολικές ε, ρυθμίσεις δεν λύνουν το πρόβλημα. Και τώρα όσον αφορά το άρθρο 16, προστασία δεδομένων, είναι κάτι το οποίο έχουμε ε, αναφέρει στην έκθεσή μας. Χρειάζονται μεν κάποιοι περιορισμοί, για τα ευαίσθητα δεδομένα. Όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο κανονισμός αυτός ε, προορίζεται στο να εμποδίσει το ξέπλυμα χρήματος και την χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να, Δεν υπάρχει, λοιπόν, λόγος να είναι η πρόσβαση απόλυτα ανοιχτή σε όλους. Πρέπει να υπάρχουν και κανόνες και ρυθμίσεις για την προστασία των δεδομένων και πρέπει να υπάρχουν επίσης και διατάξεις στις οποίες να λαμβάνονται υπόψη οι ε, δημοσιονομικές επιπτώσεις. Τέλος να πω ότι χαίρομαι πολύ για τη μελλοντική συνεργασία με τους εσκιώδεις ε, εισηγητές και με την εισηγητριά μου και ελπίζω να έχουμε μία έκθεση με σοφροσύνη που δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέρχοπ και περνάμε στους εσκιώδεις. Κύριος Νίτρας από την ΕΚΟΝ, σκιώδης εισηγητής από το ΕΛΚ και είναι παρόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Όσοι δεν γνωρίζετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας. Σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με το προσχέδιο της γνωμοδότησης. Θα πρέπει να εξετάσουμε όμως το ζήτημα των διαδικασιών που προβλέπονται στο κανονισμό. Και αυτό γιατί το πρόβλημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος στην Ευρωζώνη έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και άρα πρέπει να ακολουθήσουμε και ιδιαίτερες διαδικασίες. Για λόγους πρόληψης μπορώ να καταλάβω γιατί έχουν εκφραστεί αυτές οι ανησυχίες, δηλαδή γιατί ε, δεν θεωρείται σκόπιμο να αποθηκεύονται πληροφορίες μόνο και μόνο για λόγους ε, πρόληψης, δεδομένου του σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες οι εγκληματικές οργανώσεις τις αξιοποιούν, θα έπρεπε και εμείς που προσπαθούμε να τις καταπολεμήσουμε, να τις αξιοποιήσουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες, θα υποβάλουμε ορισμένες τροπολογίες στην γνωμοδότηση. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι αυτή, αυτός ο κανονισμός πρέπει να ταιριάξει και να υπάρχει μια συνοχή με άλλα νομοθετήματα που προετοιμάζει αυτόν τον καιρό το Κοινοβούλιο. Για παράδειγμα, τη οδηγία περιπληρωμών πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς ως προς τους ορισμούς. Δεν ορίζεται με ακρίβεια τι συνιστά σαν συναλλαγή ή τι, τι, είναι μια πάγια εντολή. Μια πάγια εντολή είναι χρηματοοικονομική συναλλαγή υπό την έννοια αυτού του κανονισμού ή όχι. Αυτό δεν είναι σαφές. Υπάρχει ακόμα ένα ζήτημα. ο ενιαίος χώρος πληρωμών στην Ευρώπη, ο οποίος έχει διευκολύνει την ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών. Αλλά το άρθρο 5 παράγραφος 1 μου δημιουργεί κάποιες ανησυχίες. Δεν θα έπρεπε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση στην οποία οι τράπεζες να δυσκολεύονται να παρακολουθούν τις συναλλαγές για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα. Τα στοιχεία που περιγράφονται στο άρθρο αυτό ίσως δημιουργήσουν προβλήματα. Από το μία προσπαθούμε να διευκολύνουμε τις διασυνοριακές συναλλαγές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την άλλη αυτό αυξάνει την έκθεση και τον κίνδυνο για νομιμοποίηση ε, από, εσόδων από κλιματικέ δραστηριότητε. Ίσως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάποια στοιχεία στο άρθρο 5, για παράδειγμα το ονοματεπώνυμο ε, του προσώπου που ξεκίνησε τη συναλλαγή. Έχω μιλήσει με ε, τραπεζικούς. Και το συμπέρασμα που έβγαλα είναι ότι χρειάζεται να συζητήσουμε περισσότερο με τον κλάδο. Γιατί κάποια από, κάποιες από τις ε, ρυθμίσεις που εξετάζουμε θα δημιουργήσουν προβλήματα στις τράπεζες. Δεν πρέπει όλες τις συναλλαγές να τις ε, βάζουμε στο, στο ίδιο τσουβάλι. Υπάρχουν διαφορές. Τώρα, έχω επίσης αμφιβολίες ως προς τον ορισμό του μεσάζοντα. Ίσως είναι υπερβολικά ευρύς. Ζητούμε από την τράπεζα να ε, ελέγξει την αυθεντικότητα, την ακρίβεια των πληροφοριών. Ε, με συγχωρείτε, το ζητούμε από τους μεσάζοντες αυτό, αλλά αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Γιατί οι μεσάζοντες δεν έχουν στη διαθέσή τους τα ίδια στοιχεία που έχουν οι τράπεζες. Επίσης, οι μέγιστες κυρώσεις διαβάζουμε ότι δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι όταν δημιουργούμε ένα σύστημα κυρώσεων, το πιο σημαντικό είναι η αναλογικότητα. 10% του τζίρου είναι ένα ποσοστό το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση των μικρότερων τραπεζών. Πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Ειδικά αυτό το κατόφλι. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι αναλογικό. Αυτό το 10% εμένα μου φαίνεται υπερβολικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μέλλο που ήταν ο σκιώδης εισηγητής από τη Λίμπε για το ΕΛΚ δεν είναι παρόν. Από τους σοσιαλδημοκράτες η κυρία Μπόσκουτ έπρεπε και αυτή να φύγει. Ούτε η, κυρία Ιντφελτ από την Άλντε φτάσαμε στους πράσινους. Κύριε Γκίγκολτ, ο οποίος αντικαθιστά τον κύριο Ταβάρες. Κύριε Γκίγκολτ, έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, θα καταθέσουμε λίγες τροπολογίες, στηρίζουμε σε γενικές γραμμές την ε, έκθεση. του κυρίου Κέρκοπ που είστε εκεί πέρα, είστε μάλιστα, και της κυρίας Κλέβα. Στηρίζουμε λοιπόν τη γενική γραμμή της έκθεσης και θέλουμε να τονίσουμε σε ό,τι αφορά το έβρος και... Uh, we και τον μοναδικό αριθμό θα πρέπει να φροντίσουμε να μην μπορεί να κρύβεται η ταυτότητα, η πραγματική πίσω από εταιρικέ δομές. Θα κάνουμε και άλλες τροπολογίες, αλλά με το χρόνο καλά τα πάμε, οπότε θα δείτε σύντομα τις ε, αναλυτικές τροπολογίες. Κύριε Σαρτζεντίνη, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τους δύο εισηγητές και όλος ιδιαίτερο τον κύριο Κίρκοπ που επέμεινε στην προστασία των δεδομένων φροντίζεται να είναι περιορισμένη η χρήση των δεδομένων να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς λόγους. Για παράδειγμα, πολύ προσεκτικά θα προσπαθήσω να δω μήπως καταφέρω να βελτιώσω, αν αυτό είναι δυνατόν, την έκθεσή σας για να ευθυγραμμίσετε με τις δικές μας προτάσεις, αλλά ειλικρινά σας ευχαριστώ γιατί πάρα πολύ καλά το διεκπαιρεώσατε το θέμα αυτό και το συμπεριλάβετε στην έκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος έχει σειρά τώρα? Ο κύριος Στρέσεκ. Δεν είναι εδώ όμως κι αυτός από την ομάδα ECR κύριος Κλούτε από την ΚΟΕ επίσης απουσιάζει. Η Κομισιόν μας είπε ότι δεν θέλει να μιλήσει. Να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος βουλευτής που θέλει το λόγο. Δεν βλέπω κανέναν. Να σας πω λοιπόν για τις προθεσμίες κατάστροπολογιών σας προτείνουμε ένα σύντομο, μια σύντομη προθεσμία, σχετικά σύντομη, επειδή είναι φιλόδοξοι οι συνεισηγητές μας και θέλουν να, να ψηφίσουμε στην τρέχουσα κοινοβουλευτική φοιτεία. Έχουν εξετάσει πολύ προσεκτικά το θέμα. Εννέα μήνες το έχουμε εδώ στο Κοινοβούλιο, άρα φαντάζομαι ότι όποιος ενδιαφέρεται είχε χρόνο να ενημερωθεί σχετικά. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι ακόμη και αν οι βουλευτές έχουν ήδη καταθέσει τροπολογίες τον Ιούλιο, αυτές οι τροπολογίες επειδή άλλαξε τη δικασία ακυρώθηκαν. Άρα θα πρέπει να επανακατατεθούν. Και για τις δύο εκθέσεις οι τροπολογίες πριν την 5η Δεκεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι. Καταλάβατε καλά τι σας είπα. Θέλει κάποιος το λόγο. Όχι. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και σας εύχομαι καλό απόγευμα και καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα από τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ να μείνουν, γιατί θα συνεχίσουμε με την προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Dear colleague, let's continue. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίσουμε. Η κατάσταση των ανθρωπινών δικαιωμάτων στην Ευρώπη το 2012, τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξής μας για σήμερα. Η συγγετής είναι ο κύριος Λουί Μισελ. Ο κύριος Μισελ παρουσίασε το σχέδιο έκθεσης στις 3 Οκτωβρίου. Είχαμε μια κρόαση στις 5 Νοεμβρίου. στην οποία ήταν παρόντες ε, οι πρόσωποι των ε, Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και της Κοινωνίας των Πολιτών και η έκθεση έλαβε 300... Ε, για την έκθεση υποβλήθηκαν 371 τροπολογίες. Θα ακούσουμε τώρα τον εισηγητή, κύριο Μισελ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συναδέλφους που συνεισέφεραν τις τροπολογίες τους 371 τροπολογίες κατατέθηκαν. Αυτό δείχνει ότι προσέχετε το θέμα αυτό και αναγνωρίζετε τη σημασία αυτής της έκθεσης για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται οι μεταφράσεις. Ε, λαμβάνω με αυτή τη στιγμή ε, τις διάφορες εκδοχές, αλλά μέχρι στιγμής δυστυχώ έχουμε τις ε, τροπολογίες μόνο στα αγγλικά. Πολύ σύντομα θα έχουμε και στις άλλες γλώσσες τροπολογίες. Την ώρα που μιλάμε έρχονται. Θέλω να εξετάσω τις τροπολογίες και να συντάξω συμβαστικές τροπολογίες, τις οποίες θα σας καταθέσω τις επόμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε που κατατέθηκαν, να σα πω ότι ω εισηγητή προτείνω σε όλου του σκιώδει εισηγητέ 70 περίπου τροπολογίε. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, ότι χρειάστηκε να περιορίσω το σώμα τη έκθεση, γιατί υπάρχουν περιορισμοί σχετικά και έτσι υπομορφήν τροπολογιών μαζί με του σκιώδει εισηγητέ που δέχθηκαν να συνυπογράψουν και πήρα και θετικέ απαντήσει από του σοσιαλδημοκράτε, του πράσινου και την ΚΟΕ χωρίς να λάβω όμω απάντηση από τους άλλους σκιώδεις εισηγητέ. Και κατέθεσα ένα πακέτο τροπολογιών λοιπόν για τα δικαιώματα των ε, ΛΟΑΔ, τα οποία συνυπογράφουν ε, οι εισηγητέ των ομάδων που σας ανέφερα και από τα μέλη του Intergroup ε, ΛΟΑΔ. Επίσης έχω καταθέσει τροπολογίες για τα άτομα με αναπηρία. Ελπίζω να στηρίξετε τις τροπολογίες αυτές το ίδιο έχουν πράξει άλλοι βουλευτές, επομένως ε, δεν πιστεύω να έχουμε πρόβλημα και θα καταλήξουμε σε συμβιβασμό που θα στηρίξουν όλοι οι βουλευτές. Έχουμε και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων. Επίσης κατατέθηκαν τροπολογίες για τα δικαιώματα των γυναικών, την εισόδα των δύο φύλων, για τα δικαιώματα των παιδιών, και θα μπορούσαμε εδώ να επεξεργαστούμε όλες τις πολιτικές ομάδες ε, συμβιβαστικές προτάσεις, ε, περιμένοντας και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Γυναικών και Ισότητας ε, Ευκαιριών. Επίσης, θα προτείνω συμβιβαστικές προτάσεις σε όλες τις παραγράφους, για όλες τις παραγράφους της έκθεσης που στις οποίες υποβλήθηκαν τροπολογίες. Δεν έχω πρόβλημα με τις περισσότερες τροπολογίες. Ελπίζω να στηρίξετε αυτές τις προτάσεις, ιδίω για τις μειονότητες ε, και συγκεκριμένα του Ρωμά, παράγραφος 17, ρατσισμός, ξενοφοβία, αντισημιτισμός και ομοφοβία, παράγραφος 18 μεταξύ άλλων. Όπου είναι δυνατόν θα προτείνω συμβαστικές προτάσεις που ελπίζω η ευρύτατη πλειοψηφία της Επιτροπής Λίμπε να τις δεχθεί. Βέβαια, το του λεχθέντος δύσκολα θα ικανοποιήσω τους πάντες. Η έκθεση εμπνέεται και διαπνέεται από την ανάγκη να λάβουμε υπόψη τις προτάσεις ε, των Επιτρόπων Παρόζο και Ρέντινγκ για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επί της ουσίας βασίζεται στην αναγνώριση του να υπάρξει ένας αντικειμενικός ουδέτερος και μη πολιτικοποιημένος μηχανισμός, ένας νέος μηχανισμός δηλαδή σε σχέση με αυτό που έχουμε μέχρι τώρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υιοθετήσει δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι στα κράτη-μέλη ή σε κράτα οποία... Ε, και έχουμε ακούσει και διάφορα σχόλια από διάφορα κράτη-μέλη. Θα κυρία Μπάουρη, κυρία Ματιέ από το ΕΛ, κυρία Ζαμπόρσκα, ο κύριος Κουρία, κυρία Σάια. Έχουν κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Προτείνουν με την παράγραφο 7, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, να διαγραφεί δική μου πρόταση, ε, διαγραφεί λοιπόν σε ό,τι αφορά την κατάσταση της Ένωσης, την ε, ομιλία του κ. Μπαρόζο το 2013 και την ομιλία της κ. Ρέντινγκ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κράτο δικαίου, αυτά δηλαδή, η τροπολογία που λέει διαγραφή ε, της επιστολής των υπουργών εξωτερικών που ζητά ένα νέο μηχανισμό αναφοράς ε, εκεί αυτό που λέμε είναι μάλλον ένα πραγματικό περιστατικό. Δεν ε, ζητάμε κάτι. Θέλουμε να διαγραφεί και αυτό. Ε, άρνηση πραγματικότητα είναι αυτό. Ε, τα είπανε ο κύριος Πάρος, η κυρία Ρέντινγκ αυτά και είναι και μέλη του ΕΛΚ να προτείνουν τώρα διαγραφή, τι να πω, επίσης για την 3 δέλτα, την παράγραφό μου και εκεί διαγραφή προτείνουν για τη συνεργασία ε, με το Συμβούλιο Ευρώπης. 3 ε για την προστασία των των δικαιωμάτων, το μηχανισμό το σχετικό, διαγραφή και αυτό, όλες τις παραγράφους, 4 και 5 για τα ίδια θέματα, παράγραφος 6, διάλογος με τα κράτη-μέλη, 7 για τις ενδεχόμενες τροποποίησεις συνδίκης, 8 αναγνώριση των παραβιάσεων θεμελιωτών δικαιωμάτων, 9 Δημόσια ένωμη τάξη, 10 για τις πτήσεις και τις ε, μυστικές φυλακές ε, τη CIA. 10, 15, 17, 18 για το ρατσισμό ξεβουλίου να αποδυναμωθεί, 21 για τη διαφάνεια, 22 για την ελευθερία κυκλοφορίας, 23 για τη δικαιοσύνη, 24 για το πίνακα επιδόσεων, scoreboard. Εδώ τίθεται θέμα, όχι μόνο πολιτικής φιλοσοφίας, αλλά και γενικότερη θέση του ΕΛ και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα έπρεπε να μας ανησυχεί. Πώς να φτάσουμε ε, όταν υπάρχει τέτοια ριζική αντίθεση με το κείμενο σε συμβιβασμούς. Αν αυτή είναι η επίσημη θέση και την έχει σκεφτεί καλά το ΕΛΚ, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε συμβιβασμού για τι παραγράφου τι οποίε σα ανέφερα. Ή τέλο πάντων δεν είμαι εγώ διατεθειμένο να υποχωρήσω πολύ από τι θέσει μου. Να προσπαθήσουμε, εντάξει. Εγώ είμαι διατεθειμένο να το προσπαθήσω. Στην προσπάθεια, εντάξει, δεν ε, θα πω όχι αλλά θα είναι δύσκολο. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή, θέλω να βρω συμβιβασμούς, αλλά το βλέπω δύσκολο. Με τις περισσότερες τροπολογίες άλλων συναδέλφων του ΕΛΚ, όπως είναι Μακοβέη και Ζαρόκα, δεν έχω πρόβλημα, ούτε με την κούε τους Πρασίνους και τους Σοσιαλιστές. Αυτά είχα να πω, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έχω δύο μέλη στον κατάλογο μελετών και ξεκινάω την κυρία Γιάροκα. Ευχαριστώ πολύ. Να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο του που ήταν δύσκολο. Διαπιστώνω ότι τίθενται θέματα τα οποία έχει συζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων και μπορέσατε να καταδείξετε ότι υπάρχουν πολλές και διάφορες τάσεις. Μες και αναφέρετε όλες αυτές τις παραγράφους. Είναι, πρέπει να είναι σαφές, πρέπει να καταφέρουμε ο διάλογος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο διοργανικός ε, διάλογος να γίνει πολύ πιο αποτελεσματικός. Παρακολουθώντας την ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, που μας ενημερώνουν για διάφορες μελέτες που έχουν διεξάγει οι υπηρεσίες, διαπιστώνω ότι εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών, διάφορες ομάδες, πολιτικές ομάδες, πολιτικά κόμματα, αλλά και ε, άλλοι οργανισμοί, άλλοι φορείς προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ως εργαλείο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μέσω της έκθεσής σας να δώσουμε μια πιο αντικειμενική παρουσίαση των θεμάτων αυτών. Παλαγμένη από τέτοιου τύπου σκοπιμότητες, γιατί θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα φέτος, που είναι ε, χρονιά εκλογών. Γιατί δεν πρέπει να ε, εγκαταλείψουμε και να απογοητεύσουμε τους ψηφοφόρους μας στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Γι' αυτό καλωσορίζω τις παραγράφους τις οποίες αναφέρεστε σε, στα άτομα που βρίσκονται σε ε, εξαιρετική έμβια, στους φτωχού στην Ευρώπη, καθώς επίσης και τον ρατσισμό κατά τον Ρωμά ή άλλων ομάδων. Δυστυχώς τα όρια της ε, έκτασης της έκθεσης δεν μας επιτρέπουν να συμπεριλάβουμε περισσότερα οικονομικά επιχειρήματα, αλλά θα πρέπει να καλέσουμε για περισσότερη δράση και από την πλευρά της Επιτροπής και από την πλευρά των κατών μελών. Ανοίγει έτσι ένα παράθυρο μέσα από αυτή την έκθεση. Να τονίσουμε ότι στις περιοχές εκείνες, στις χώρες εκείνες που έχουν χτυπηθεί από την οικονομική κρίση και στις οποίες καταφτάνουν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια αυτά χρησιμοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και να φτάνουν τελικά στα πλέον φτωχά στρώματα της κοινωνίας. που υποτίθεται ότι εκείνα ακριβώ τα στρώματα στοχεύουν τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τονίσουμε τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ του ρατσισμού, της ξενοφοβία, του αντισημιτισμού και του ρατσισμού κατά των μεταναστών ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται να ασκήσουμε πίεση στην Επιτροπή και το Συμβούλιο για να λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές της αλληλεγγύης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις όποιες πολυόμενους μήνες. Θα πρέπει επίσης να μιλήσουμε για το ζήτημα της γετοποίησης των παιδιών των Ρωμά στα σχολεία και ελπίζω να καταλαβαίνει τη σημασία της, του θέματος η Επιτροπή. Ε, προετοιμάζεται μια μελέτη ε, για το θέμα αυτό και διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση είναι τραγική όχι μόνο στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και σε, όλες, και σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Η περιφερειοποίηση και η γετοποίηση των παιδιών των Ρωμά δεν έχει περιοριστεί, δεν έχει καταπολεμηθεί όπως θα έπρεπε. Και πρέπει να είμαστε σαφείς και να πούμε ότι αναμένουμε και απαιτούμε από την Επιτροπή να αναλάβει δράση για αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Γιάροκα. Μια και ο κύριο Κέρκοπ πρέπει να φύγει σύντομα, δίνω αμέσω τώρα στο, το λόγο σε αυτόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λυπάμαι για το ότι αυτά που θα πω δεν είναι και τόσο θετικά. Ξέρω ότι ο κύριος Λούις ε, Μισελ έχει μια σαφέστερη εικόνα της θέσης μας και δεν θέλω να είμαι αγνώμων, διότι παρά το ότι το κείμενο είναι έφτασε πρώτο στην αγγλική γλώσσα και μου επέτρεψε να το κοιτάξω πολύ καλά. Λυπάμαι ωστόσο για την αρνητική μου στάση στην έκθεση αυτή. Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο και το έχω πει πολλές φορές αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι και δικαστής ε, και κατηγορούμενος όσον αφορά το ποια κράτη παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ποια όχι. Εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχουμε υποβάλει τροπολογίες, όχι επειδή ε, νομίζουμε πως είναι τέλεια έκθεση, το, το αντίθετο. Ε, αλλά προσπαθήσαμε να υποβάλουμε μία τροπολογία να καταργηθεί, να τη γραφεί έκθεση και να γίνει έκθεση πρωτοβουλία, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό. Τώρα, ορισμένα σημεία με ενοχλούν ιδιαίτερα. Η τροπολογία 109 που αναφέρεται ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα νέο μηχανισμό τη Κοπενχάγη. Αδυνατό να συμφωνήσω με αυτό. Μετά, 103 για την διαδικασία παγώματο, όπου τα κράτη-μέλη κατόπιν μπορούν να αναστείλουν ε, νόμους όταν ε, παρεβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό παρεβιάζει την αρχή της επικουρικότητας και το θεωρώ δύσκολο και δεν ξέρω και αν είναι και νομικά ε, θεμητό. Έπειτα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο δεν έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει στις αποφάσεις ε, των κρατών μελών να επιβάλλουν στρατιωτική θητεία στους πολίτες τους και να τους τιμωρούν αν την αποφεύγουν. Δεν υπάρχει κάποια νομική βάση σε αυτό. Τέλος, πολύ φοβάμαι ότι αυτή η έκθεση, όπως και αρκετές άλλες, έχει γίνει κάτι σαν ε, χριστουγεννιάτικο δέντρο ή κάτι έχει σαν χωματερίο, όπως θέλετε πάρτε το, όπου ο καθένας μπορεί να αφήνει τις ανησυχίες του και τα διάφορα, ε, τις διάφορες επιθυμίες του, τις ε, πολιτικές. Υπάρχουν άλλα μέρη για να κάνει κανείς κάτι τέτοιο. Αυτό, σε αυτό συμπεριλαμβάνεται το κυπριακό ζήτημα, το ζήτημα της Τουρκίας, η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα και να πω ότι, παραλαμβάνω, δεν έχουν θέση αυτά μέσα στην έκθεση. Επίσης, δεν θεωρώ πως είναι σωστό ή λογικό να χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους ε, γλώσσα και διατύπωση. Η έκθεση αυτή έχει αξία όσον αφορά ε, την χρήση σαν πλατφόρμα, όμως δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε ε, για να εισαγούμε τέτοιου είδους τροπολογίες και λυπάμαι γι' αυτό. Και ξανά λυπάμαι και συζητώ συγγνώμη από τον κύριο Λουί ο οποίο είναι πραγματικά ε, άριστος τεχνίτης του λόγου, αλλά δεν μπορώ να στηρίξω την έκθεσή του με τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κέρκοπ. Κυρία Σντανόκα. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ο κύριος Κέρκοπ να ακούσει και τη δική μας άποψη και να μην φύγει αμέσως. Διότι εντάξει, σεβόμαστε το δικαίωμα να έχετε άποψη, να έχει ο καθένας μας άποψη. Εάν όμως θέλετε να είστε συνεπείς, πρέπει να απορρίψετε και όλες τις εκθέσεις και τις ε, συστάσεις ε, που σας λένε ότι δεν μπορείτε να συμπεριφέρεστε σαν να μην ανήκετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, να ψηφίζετε στις επιτροπές, στο Στρασβούργο για θέματα, για την ύφεση, και μετά να νύπτετε τα σχήρα σας. Όχι, αν θέλετε να... Αν θέλετε, αν, μάλλον όποιος ε... ζει σε ένα γυάλινο σπίτι δεν πρέπει να πετάει πέτρες. Και ε, έτσι έχουμε οδηγηθεί σε μια κατάσταση που είναι κάθε άλλο από τέλεια. Και δεν υπάρχει και πολιτική θέληση κιόλας για να γίνουν αλλαγέ προ το καλύτερο. Η δική μα ομάδα έχει στείλει επιστολή στον πρόεδρο πολλέ φορέ και όχι μόνο μία φορά για να ζητήσει να υπάρχουν ε, εκθέσει ε, χώρα. Και τέλος αυτή η προσέγγιση έτυχε ε, στήριξη από πολιτικές ομάδες, όχι από τη δικιά σας βέβαια, όχι από τους ε, συντηρητικούς. Επίσης, Μιλώ εκ μέρου της ε, κυρία Λούνατσεκ, της κοιότητας εισηγήτρια των Πρασίνων, που απουσιάζει. Και θα ήθελα να πω, η και μάλλον, ο Ρούι Βάρε και εγώ, ότι υποβάλαμε τροπολογίες στην έκθεση του κύριου Μισελ και με τις τροπολογίες αυτές θέλουμε να δηλώσουμε την εκτίμησή μας στο κείμενο να εκφράσουμε την ευχαρίστηση και την ευγνωμοσύνη μας ε, για το κείμενο αυτό. Λυπούμεθα ο, για το ότι δεν έχουμε συμβιβασμούς και συμβαστικές λύσεις να συζητήσουμε σήμερα, αλλά ελπίζουμε ωστόσο να συνεχίσουμε την ε, καλή συνεργασία Γι' αυτό λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις τροπολογίες, άρθρο 3. Συμφωνούμε πως υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των ε, συνθήκων και να υπάρχει συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης μέσω μιας ε, κοινής Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Ωστόσο, το, η πρόταση του να δημιουργηθούν ε, πίνακες ξεχωριστή και συνολική αναχώρα για την κάθε χώρα είναι κάτι που μας αρέσει ιδιαίτερα και το έχουμε προτείνει και ως ε, τροπολογία. Υπάρχουν συγκεκριμένες τροπολογίες για την πολιτική που θα ακολουθηθεί για τα θεμελιώδη δικαιώματα και πώς θα συνδεθεί αυτή με την οικονομική πολιτική και το Συμβούλιο. Ελπίζουμε να στηρίξει την πρότασή μας. Κάπως έτσι είναι το περιεχόμενο της τροπολογίας μας. Επίσης, πάλι για, την, για το άρθρο 3, προτείνουμε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αξιολόγησης ομοτήμων σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως ακριβώς ε, υπάρχει και ένας παρόμοιος μηχανισμός στον ΩΣΑ. Τώρα, σχετικά με την παράγραφο 4, όπου γίνεται λόγος για τον νέο αυτό μηχανισμό για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την ε, των αξιών της Ένωσης που ε, αναφέρεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης και της Χάρτας των ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Να προσθέσουμε και κάποιες δικές μας ιδέες για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένας τέτοιος μηχανισμός. Για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει μια οριζόντια προσέγγιση Ε, στοιχεία συντονισμού, συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Και πλήρη συνεργασία όσον αφορά τις ε, παραβιάσεις των ε, διατάξεων του άρθρου 2. Καθώς επίσης και αναφορά στο σημείο F όπου αναφέρεται αυτή η διαδικασία παγώματος σε περίπτωση τέτοιας διαδικασίας η Κομισιόν θα διεξάγει έκτακτες συνεδριάσεις με τα κράτη-μέλη και τα λοιπά και τα λοιπά. Πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 2 και διασφάλιση αυτής. Επίσης υποβάλαμε κάποιες τροπολογίες για την ε, συνέχεια της παρακολούθησης ε, και της εφαρμογής αυτής. Προτείνουμε μια νέα παράγραφο 6α. Επίσης, μια νέα παράγραφο 15α. όπου αφορά τους ε, νέους ανθρώπους που κατηγορούνται και φυλακίζονται ε, επειδή είναι αντιρρησία συνείδησης της στρατιωτικής θητείας. Και πιστεύουμε ότι αυτά τα στοιχεία αξίζει να αναφερθούν και πρέπει να αναφερθούν επίσης. Υπάρχει και ε, ένα πρόβλημα, το πρόβλημα των απάτριδων σε μεγάλους ε, αριθμούς αυτή. Η κατάσταση και το αυτό φαινόμενο είναι πάρα πολύ έντονο στη χώρα μου και στην Εστονία. Εμείς λοιπόν έχουμε υποβάλει μια πρόταση που υπάρχει και, στην και σε μια προηγούμενη έκθεση όπου οι απάτριδες οι οποίοι όμως ε, μένουν, διαμένουν μόνιμα σε ένα κράτος ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνουν το δικαίωμα ψήφου. Επίσης, προτείνουμε μία νέα παράγραφο 22α και μία παράγραφο 24α, επίσης καινούρια, όπου θα προβλέπεται αξιολόγηση του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη. σας έχουμε διανέμει το σχετικό κείμενο. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω σε ε, συνέχεια της συνεργασίας μας και σε εφαρμογή και συμπερίληψη των προτάσεών μας και των συμβιβαστικών τροπολογιών στο κείμενο. Ξανά, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μισελ και καλή τύχη. Ευχαριστούμε. Κυρία Γκίνκα Γκέτς, ευχαριστώ πολύ. Λυπούμε που έφυγε ο Σκύρκοπ. Πριν ακούσει τη δική μου άποψη. Που φυσικά δεν θα σας εκπλήσει, διαφέρει πολύ από τη δική του. Για την έκθεση πάντα. Βέβαια τη συζήτησή μας θα τη συζητήσουμε, θα τη συνεχίσουμε όταν συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες για αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Πολλές φορές έχουμε πει ότι εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, είμαστε πολύ καλοί όταν πρέπει να προστατεύουμε τους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς μας κανόνες, αλλά πολύ πιο αδύναμοι σε ό,τι αφορά τι θεμελιώδεις αξίες. Αυτό το οποίο εκτιμώ όλο ιδιαίτερο στην έκθεση αυτή είναι ότι ο Λουί Μισελ προσπαθεί να προωθήσει τις ε, πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν με την έκθεση Ταβάρες και με τους υπουργούς εξωτερικών και η Κομισιόν υποσχέθηκε ότι θα ε, δημοσιεύσει ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Πρωτοβουλίες λοιπόν που μιλούν για τις ε, αναγκαίες μεθόδους και τρόπους για να προστατεύσουμε σε μελιώδες μας αξίες, κράτος δικαίου, δημοκρατία, και όλα τα άλλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες που είναι σε κίνδυνο. Η κρίση βλέπουμε ότι υπονομεύει τις θεμελιώδεις αυτές αξίες, βλέπουμε όλο και πιο ακραία εξτρεμιστικά κόμματα να αναδύονται, που αμφισβητούν αυτές τις θεμελιώδεις αξίες, αλλά την τάση αυτή βλέπουμε ότι να ακολουθούν και τα πιο ε, mainstream κόμματα. Ο Λί Μισελ στο πιο σημαντικό κομμάτι της έκθεσης του προσπαθεί να συμπεριλάβει τις ε, δυνατότητες που μας δίνουν ε, οι συνθήκες για το τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα και τι είδους αλλαγές, ε, τροποποιήσεις των συνθήκων ενδεχομένως χρειαστούν στο μέλλον. Γιατί αυτά πρέπει να τα προετοιμάσουμε ενδεχομένως. Δεν είναι μια δεδομένη πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και πολλές άλλες πτυχές, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες της έκθεσης και ελπίζω πραγματικά να υποστηριχθεί από μια ισχυρότατη πλειοψηφία. Συμφωνώ και με ένα μεγάλο μέρος των τροπολογιών για την κατάσταση των μειονοτήτων, για τους Ρωμά, αύξηση ξενοφοβίας, ε, αντισημιτισμού κτλ. Έχω καταθέσει και εγώ τροπολογίες για τα θέματα αυτά, αλλά νομίζω ότι πέραν των τροπολογιών αυτών θα πρέπει το βασικό μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα της έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας να διατηρηθεί, ελπίζοντας να στηριχθεί, όπως είπα, από ευρύτατη πλειοψηφία. Βερζιά. Excusez-moi. Euh, et excusez également mon, mon retard. Συγγνώμη που έβηξα και συγγνώμη που έφτασα και καθυστερημένη. Δεν άκουσα ε, τον εισηγητή, ε, τον οποίο όμως θέλω να ευχαριστήσω παρόλα αυτά για την ε, έκθεση που προετοίμασε λαμβάνοντας υπόψη να το δυνατόν περισσότερο τους σκιώδες εισηγητές. νομίζω ότι διεπόμαστε από την κοινή λογική, την δική του, την προσέγγιση δηλαδή. Υπάρχει βέβαια ένα φιλοσοφικό ζήτημα προσέγγισης ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων που ξύνεται θα έλεγα. Η λογική της συνθήκης της Λισαβόνας. Ήμουν ε, αντίθετη, ήμουν πολέμη, αλλά τέλος πάντων υπάρχει πλέον και πρέπει να την αξιοποιήσουμε στον το περισσότερο. Ήταν ότι συμπεριέλαβε το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι το θέμα αυτό που μας ε, απασχολεί. Είτε συμφωνούμε με αυτή την ε, ιδέα της συμπερίληψης των ε, θεμελιών δικαιωμάτων και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή πρόοδο, και νομίζω ότι αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε στην Επιτροπή μας από την αρχή αυτής της θητείας, ιδίω φάση της πρώτης έκθεσης που καταρτίστηκε τη δική σας, κυρία Γκάλ. Είτε προσπαθούμε Μπορούμε τις δυνάμεις να αποφύγουμε την ε, πρόοδο σε αυτό το θέμα. Και αυτές τις δύο λογικές τις βλέπουμε ε, να διαγωνίζονται στην Επιτροπή αυτή, αν δει και τον αριθμό των ε, προτάσεων διαγραφής. Εγώ θα ήθελα να δώσουμε μια οικουμενική ε, διάσταση. Έχουμε την οικονομική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών και τα κράτη-μέλη έχουν προσχωρήσει σε αυτήν την οικουμενική διακήρυξη. Μήπως δεν είναι τελικά κάποιοι σύμφωνοι πλέον με αυτή τη λογική. Θα ήταν καλύτερο να το πούμε αυτό. Εγώ συνεχίζω να βλέπουμε αυτή τη λογική και θεωρώ ότι είναι κατεπήγον να δράσουμε για κάποια ζητήματα και ιδίω πάνω σε αυτά έχω καταθέσει και κάποιες τροπολογίες συγκεκριμένο. Να καταπολεμήσουμε την άνοδο του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και να καταπολεμήσουμε και όλες τις διακρίσεις που βλέπουμε να επανεμφανίζονται δυστυχώς. Επέμεινα επίσης στο θέμα της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Στην αρχή της θητείας είχαμε ακούσει ότι θα ήταν θέμα εβδομάδων μηνών και φτάνουμε στο τέλος τώρα της θητείας και δεν έχουμε προχωρήσει. σε μικρό σημείο και από πίσω έχουμε τη δυσκολία επικύρωσης, πίσω μάλλον από τη δυσκολία αυτής της επικύρωσης έχουμε ιδεολογικές μάχες. Αυτή τη φιλοσοφική θεώρηση, όπως σας είπα, για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αρνητική θεώρηση των πραγμάτων. Με όλα αυτά δεν θα καταλάβει μεγαλύτερο χώρο στο παγκόσμιο προσκήνιο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πέμπτη απόγευμα δύσκολα μπορεί κανείς να μιλήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν βλέπουμε να καταπατώνται και στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εντάξει, τώρα στο κατά πόσο γίνεται στον ίδιο βαθμό με άλλες περιοχές του κόσμου είναι υποσυζήτηση. Κύριος Μισελ. Ευχαριστώ. Οι περισσότεροι από τους προλαλήσαντες στην πραγματικότητα απάντησαν αυτά που ήθελα να πω κι εγώ σε εκείνους που διαφωνούν με την εκθέσή μου. Πράγματι, υπάρχει ένα πρόβλημα φιλοσοφικής φύσεως. Δεν μπορούμε να θεωρούμε. Απ' τη μία, ότι εντάσσουμε το χάρ, τη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη συνθήκη αυτή η Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι το σημείο αναφοράς με βάση το οποίο θα έπρεπε να κρίνουμε την κατάσταση στις διάφορες χώρες και μετά την άλλη όπως έκανε η κυρία Τάνοκα να προσπαθούμε συνέχεια να επικαλεστούμε την αρχή τη επικουρικότητας για να αποφύγουμε να αναδείξουμε και να αποφύγουμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Τι είπατε? Ε, συγγνώμη, όχι κυρία Ζδάνοκα, ο κύριο Κέρκοπ το είπε αυτό. Τι είπα και εγώ. Αυτός ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να αποφύγουμε, να σεβαστούμε μια συνθήκη την οποία έχουμε προσυπογράψει ε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αρχή της επικουρικότητας για να καταπολεμήσουμε οτιδήποτε δεν αρέσει στις εθνικές κυβερνήσεις. Το κεκτημένο της συνθήκης, οι προηγούμενες εκθέσεις που έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώ επίση και σχετικέ δράσει τη Επιτροπή, προφανώ είναι σημείο αναφορά. Εάν δεν βασιζόμαστε σε αυτά, σε τι θα βασιστούμε. Ε, διαφορετικά, α το πούμε ανοιχτά, όπω είπατε και εσεί συνάδελφε, προηγουμένω, α πούμε ανοιχτά ότι πλέον δεν μα ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν θέλουμε να τα σεβόμαστε. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αποτελούν αξία την οποία μας, ε, που μα αφορά, τα αγνοούμε δεν τα σεβόμαστε, δεν έχουν πλέον νομική αξία, δεν έχουν πλέον θεσμική αξία ε, κτλ. κτλ. Αν κάποιοι άνθρωποι καιροσκόποι σκέπτονται έτσι, δεν μπορώ εγώ να τους ε, σταματήσω. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση αξιών. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε μηχανισμούς και συστήματα που εξετάζουν κατά πόσο τηρούμε αυτές τις αξίες μου θέτουν το ερώτημα για παράδειγμα της θεσμικής νομιμοποίησης του έργου μας, του κοινοβουλίου μας. Ε, δεν είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαρνηθεί το δικαίωμα του να εκφράζει άποψη επί των θεμάτων αυτών. Ίσως εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση και πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Μου λένε. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι την κριτική, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η έκθεση μου λένε η χρησιμοποιεί τα ανθρώπινα δικαιώματα ως εργαλείο πολιτικής. Όχι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Κάνουν αυτοί που επικαλούνται την αρχή της επικουρικότητας με τρόπο ε, ε, τέτοιο σοκαριστικό να επικαλούνται αυτήν την αρχή για πολιτικές σκοπιμότητες. Είτε σεβόμαστε τη χάτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε όχι. Απλό είναι το θέμα. Είναι απλό να κρίνουμε εάν ένα κράτος σέβεται ή όχι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη θα αρχίσουν να ανακύπτουν όλο και περισσότερα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να ε, συνέχεια να εφιστούμε την προσοχή του, του κοινού στο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται στις χώρες ΑΚΕ ή στην Ασία, στην Αφρική και τα του οίκου μας να μην μπορούμε να τα αγγίξουμε εγώ όπως σας είπα θέλω να προσπαθήσω να βρω συμβιβαστικές λύσεις. Αλλά όχι και μέχρι το σημείο του να τα ξεπουλήσω όλα, υπάρχουν και όρια. Εάν βλέπω αυτή την προσέγγιση από την απέναντι πλευρά και εγώ θα γίνω πιο ε, αυστηρός. Θα σκληρύνω τη στάση μου. Αν μου ζητούν τελικά να πουλήσω την ψυχή μου στο διάβολο για να έχουμε συμβιβαστική λύση, όχι. Δεν πρόκειται να το κάνω. Γιατί υπάρχει μία πτυχή αυτού του ζητήματος που είναι σημαντική. Και έχετε δίκιο, κύριε συνάδελφε, το ζήτημα το οικονομικό. Δεν είναι δυνατό να, μην πούμε ότι η οικονομική κρίση έχει αρνητικό αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως σας είπα λοιπόν, θα κάνω ό,τι μπορώ για να βρούμε συμβαστικές, αλλά χωρίς να χάσουμε και την αξιοπρέπεια μας. Πραγματικά δεν θέλω καυγά να κάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά κάποιες από τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί στην πραγματικότητα προσπαθούν να υπονομεύσουν την ουσία της έκθεσης, όχι μόνο της έκθεσης, την ουσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και με συγχωρείτε από τη συνάδελφη, αλλά προφανώς όσοι καταθέτουν τέτοιες τροπολογίες δεν αναζητούν συμβιβασμό, απλώς θέλουν να προκαλέσουν θόρυβο που δεν έχει καμία σχέση με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ίσως για λόγους πολιτικούς ή φιλοσοφικούς που αδυνατό να καταλάβω. Πρέπει να σεβαστούμε και το πνεύμα και το γράμμα των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει. Διαφορετικά Καταλαβαίνουμε γιατί ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πλέον την, αυτή την υποκρισία στην Ευρώπη. Και εν πάση περιπτώσει εγώ δεν σκοπεύω να συμμετάσχω σε τέτοιου τύπου υποκρισία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μισελ. Πρωτού ολοκληρώσουμε την απογευματινή συνεδρίαση, πρέπει να σας πω ότι η ψηφοφορία για την έκθεση θα διεξαχθεί στην Επιτροπή ΛΥΠΕ στις 16-17 Δεκεμβρίου και η επόμενη συνεδρίαση μας ε, θα έχει τη μορφή Διερευνητικής Επιτροπής στις 2 Δεκεμβρίου από τις 3 έως τις 6.30 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και καλό βράδυ να έχετε.